ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ανακοινώσεις της Προέδρου, τις αποφάσεις των συντονιστών στην ε, χθεσινή συνεδρίαση 9 Ιουλίου. Θα τις βρείτε, όπως έχουν μοιραστεί, και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις έως τις 12.30 θα, θα θεωρηθούν εγκεκριμένες. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας με τις ψηφοφορίες. Και να ξεκινήσουμε για να δούμε ότι είμαστε όλοι εδώ. Αρχίζουμε. Πέρας. Πολύ καλά. Κύριε Βαντακάμ, τελειτουργεί λειτουργεί η κάρτα σας. Ο Ισμαήλ Ερτούγκ είναι εκεί για να σας βοηθάει όμως. Πάμε. Ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Κριστίν Ριβό Νταλόν για τους ε, κοινούς κανόνες, μάλλον για τα καινούργια επιβετικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά ε, οχήματα ε, της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Ξεκινάμε, είστε έτοιμοι. Πάμε. 140 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε ε, έλεγχο να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπάρχει κάποιος παραπάνω σε κάποια ομάδα. Κάποιος θα πρέπει να μην ψηφίσει. Για να επαληθεύσουμε, πέρα της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Α, δεν έχετε την κάρτα σας μαζί. Και τι ψηφίσατε. Υπέρ. Δεν αλλάζει όμως και τίποτα. Δυστυχώς. Απορρίπτεται. Θα πρέπει να μας δείχνετε κάθε φορά τι ψηφίζετε όμως. Θα σας κοιτάζω. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 142, 25, 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Θέλετε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Και συνένας γιατί ε, η συνάδελφος δεν έχει την κάρτα της. Πέρας. Δεν απορρίπτεται, διότι ε, η συνάδελφος δεν έχει την κάρτα της, ψηφίζει υπέρ. Άρα εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την 143. Μία ψήφος κατά επιπλέον. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με μία ψήφο επιπλέον. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι πολύ μικρή διαφορά να αληθεύσουμε Έχουμε και μία ψήφο παραπάνω κατά. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Συμβιβαστική 2α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2B, 2Β, b υπερ κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός, 2B. Πέρας, εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα. Τροπολογία 170. 170. Κύριε Βαντενκάπ, το βρήκατε. Γυρίστε σελίδα. 170. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Θα το επαληθεύσουμε. 31. Έχουμε μία ψήφο παραπάνω τόσο ή άλλως. Πέρας. Απορρίπτεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 ταυτόσημες. 32. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά Ναι κύριε Ρεβονταλόν θέλετε να ξαναψηφίσουμε Όχι μπορούν να ψηφιστούν 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Ελέγχουμε. 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ταυτόσιμες 33-176. Υπέρ. Κατά εποχες απορριπτονται απορρίπτονται. Δύο ταυτόσιμες πάλι 34-177 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 180 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 182. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τι ψηφίσατε εσείς. Οπότε εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Κόχ που τα προσέχετε όλα. 183, 84, 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τρεις ταυτόσιμες. 186, 187, 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Εγκρίνονται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτει. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Εντάξει. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά κύριε Κονταλόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την 189. Πέρας. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε δεν με πιστεύεστε. Εντάξει λοιπόν, 190. Πέρας. Απορρίπτεται. Ταυτόσιμες 191-92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται νομίζω, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 191-92. Πέρας. Εγκρίνονται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. απόχέ, Αποχές. Απορρίπτεται. ταυτοσιμε ταυτόσημες 38-195 υπέρ. Κατά. αποχέ Να επαληθεύσουμε. Γιατί δεν ειναι σαφε σαφές. 38-195. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τρία Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε, οπότε θα ψηφίσουμε μία-μία όλες τις τροπολογίες. 196, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε την 197. Πάμε. Το αλέλε μπλε είναι το βράδυ. Πέρας. Απορρίπτεται. 40. Να συνεχίσουμε. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για την 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Εντάξει, να ελέγξουμε για τη 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 200 απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207 Καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκε 206, συγγνώμη. 43, 208 και 209. Δεν διάβασα σωστά, με συγχωρείτε. Συμβαστική 5 απευθεία. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύο ταυτόσημες 218-219 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας για αυτές τις δύο εγκρίνονται. 220, 221 μάλλον, 222 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Για να ελέγξουμε. 224. Πέρας. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε διότι δεν λειτουργήσε το μηχάνημα. Ξανά. 224. Πέρας. Απορρίβεται. 225 υπέρ. Κατά. Έχετε κουραστεί, ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να με εμπιστεύεστε κύριε Ρικέ. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 228-229 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 230. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε. Πέρας. Η συμβαστική 6 απορρίπτεται. Καλά δεν έκανα που έλεγξα. 147 Μάλλον 47 εγκρίνεται. 47 επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Ταυτόσιμες. 48-233. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 234 του κυρίου Έκχαουτ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ταυτόσιμες, 49-235, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Αλλά πρέπει και να το απαλληθεύσουμε 49 και 235, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 238 υπέρ. Κατά. Κύριε Βάντεν δεν καταλαβαίνω γιατί καταψηφίζετε τις δικές σας τροπολογίες κάθε φορά. Κάποιες φορές πραγματικά, τι να σας πω, Απορρίπτεται νομίζω. Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή κάποια φορά. 240 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Αλλά να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε και την ε, συμβαστική 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Α, καταπίπτει αν εγκριθούν οι προηγούμενες. 50. 50 υπέρ. Ποιο είπε όχι, όχι. Κυρία Γιούτο, τι θέλετε. Μόλις 9.28 είναι η ώρα. Εντάξει, κυρία Γιούτο, να συνεχίσουμε. 50 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 50. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι επαληθεύουμε την 52 λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 240 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 κατά εποχές επαληθεύουμε την 54 Πολύ θορυβόδηση είναι η Κομισιόν σήμερα. Τι συμβαίνει. Λήξη ουφορίας; εγκρίνεται. 2.59 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση έναρξη της ψηφοφορίας λήξη απορρίπτεται 256 και 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε. Εγκρίνεται. Ήταν ταυτόσιμες αυτές οι δύο τροπολογίες. Περνάμε στη 258. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτεται. 263. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 264. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 265. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Mm. Όλες οι τροπολογίες επόμενης σελίδας καταπίπτουν εξαιτίας του συμβιβασμού 1β. Περνάμε κατευθείαν στην 287. 287, 288 και 289 που είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε. λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.92 υπέρ. 2.92. Κανείς δεν υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 2,90 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 2,91 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 2,93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,94 υπέρ. Κατά Εποχές Δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2,95 και 2,96 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Και εδώ επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τι θα πει προφανώς. Συνεχίζουμε. 297-298 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ Συγγνώμη, 301 λέει πρόεδρο. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Δύο τροπολογίε. Όχι, καταπίπτει. 304, 305, 380 και 306. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές επαληθεύουμε την 308. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 309 και 311 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τρία δώδεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 3.13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.14 και 3.15 υπέρ. Είναι ταυτόσιμες. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 3.16 και 3.17 καταπίπτουν. Και όλες μέχρι

εποχές εγκρίνονται 334, 335 και 336 υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται μετά καταπίπτουν 357. Τι λέτε? 357. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 358 και 359 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 361 κατά πίπτη. 360 επίσης. 362 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 363, 64 και 65 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 και 3, 366 και 367 υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτονται. Ξήντα τρία. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται δυστυχώς. 368 υπέρ Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 369 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 370 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 371 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. 3.72, 3.84, 3.73. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτονται. 3.74. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 3.75 και 3.76 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνονται. 3.77 υπέρ. Κατά αποχές απολύπτεται. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. 3.78-3.79 υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνονται. Περνάμε στην αιτιολογική έκθεση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαληθεύουμε. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Για την 66 λέω. Η 1 εγκρίθηκε. Η 67 και η 68 καταπίπτουν. Οπότε περνάμε στην 66. Ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Επαληθεύουμε την 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη πληροφορία. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75, υπέρ, κατά, Εποχές, Δεν ξέρω τι γίνεται. Επαλήθευση. Τις 75. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 καταπίπτει. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 80. Ένα εξωφορίας. Εγκρίθηκε, μπράβο. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας το επαληθεύσουμε όμως. Τροπολογία υπερθυμών 5. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας το δούμε. Συμβαστική υπαριθμόν 9. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται πράγματι. 8. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ. Non, non, il y a une erreur, il écrit euh, Έγινε ε, ένα λάθος εδώ, δεν είναι 88, είναι 89, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Όλα είναι υπό έλεγχο. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 90. Καταπίπτει. Θέλετε να επαληθεύσουμε τη 10. Ωραία. Βεβαιώνουμε, επαληθεύουμε τη 10. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη. Φοράτε ακουστικά και μιλάτε πολύ δυνατά. Απορρίπτεται η 10. Ευχαριστούμε κύριε Κόρ. Περνάμε στην 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να το επαληθεύσουμε. Οκ. Okay. 90. Λήξη ουσφορίας. Με ρωτάτε τι κάνω. Σας κοιτάω. Εσείς δεν κάνετε κάτι, δεν σηκώνετε το χέρι σας. Σηκώνετε λίγο το χέρι σας. Εγκρίνετε 90. 91. Όχι, καταπίπτει. Κύριε Βερκόνεν, πολύ δυνατά μιλάτε. Σας παρακαλώ πολύ. Βγάλτε λίγο τα ακουστικά σας και θα είτε θα μιλάτε λιγότερο δυνατά. 91. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Οχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες ε, υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτονται 96 και 97. 12, 98 και 99 και πάλι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά εποχές Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 105 και 106 ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσιμες 14 και 107 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 108 και 109 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 και 112 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 19. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Συγγνώμη. 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουν ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου άρχεται η ψηφοφορία Λίγη. «23 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται». Έχει το λόγο η συγκήτρια. Θέλω να διαγραφεί το όνομά μου από την έκθεση. Να αποσυρθεί. Λαμβάνω υπόψη και καταγράφουμε το αίτημά σας. Σημειώνετε στα πρακτικά το αίτημά σας. Να συνεχίσουμε παρακαλώ. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καναδά για τις αεροπορικές μεταφορές. Περνάμε απευθεία στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Εάν θέλετε να βγείτε, ησύχως παρακαλώ. Ψηφίζουμε τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καναδά. Απευθείας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. 39 υπέρ, μία ψήφος κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται η εντολή. Και τώρα δεύτερη ψηφοφορία για το πρωτόκολλο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Καναδά. Λόγω και της προσχώρησης της Κροατίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Κροατία. Το βρήκατε. Κύριε Κράμερ, το πρωτόκολλο ψηφίζουμε. για να μπορέσει και η Κροατία να προσχωρήσει στη σύμβαση, στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καναδά. Πέρα τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε. Αγιούτο. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο. Ε, υπάρχουν ψηφοφορίες σε διαφορετικές ε, επιτροπές, ε, οπότε ίσως ε, θα μπορούσαμε, χωρίς να αναφέρετε τα amendments, να προχωρούμε γρήγορα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, θα πρέπει να πάμε στις άλλες επιτροπές για τις ψηφοφορίες, οπότε να μην λέτε amendment τα κάθε φορά, να λέτε κατευθείαν το νούμερο. Donc on va être sur votre volet, madame. Θα ακολουθήσουμε την επιταγή σας, κυρία Μάισνερ. Ωραία λοιπόν, μόνο νούμερα για να κάνουμε γρήγορα. Συμβαστική 1, έκθεση Αγιούτο. 1, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προστίκη στην συμβαστική 2, για την προστίκη, υπέρ, είναι από κάτω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Κάνετε πολύ θόρυβο και στο βάθος. Εάν θέλετε να μιλήσετε έξω. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την προστίκη για τη συμβαστική 2. Τη βρήκατε όλοι. Προστίκη. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τότε γιατί φωνάζετε τσεκ. 150. Εάν ο καθένα μιλάει, δεν θα τα καταφέρουμε. Αποφασίσαμε να λέμε μόνο του αριθμού χωρί να λέμε και τροπολογία. Παρακαλώ να παρακολουθείτε. 157 απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 16 και 165. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική ψηφοφορία και οι δύο. 16 και 165. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169. Υπέρ. Α, δεν ψηφίζεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Καταπίπτει 175. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 79 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 179. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 180. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 182. περ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απευθείας στην 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε απευθείας στην 193 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100... Απευθείας 209. Θέλετε έλεγχο για την 196. 196 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απευθείας 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πανομοιότυπες 25-221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται έλεγχος 25-221 ταυτόσημες. 25-221. Πέρας. Εγκρίνονται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 224 υπέρ. Με συγχωρείτε. Πάμε απευθείας στην 27. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 227 καταπίπτει. 28 ένβη. Υπέρ. Α, και αυτή καταπίπτει. Με συγχωρείτε. 27 μάλλον. Ένβη 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ. Ψηφίζουμε την 228. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 229. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Θέλετε έλεγχο. Ελέγχουμε για τον 229. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 32. Άρχια την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δίκιο είχατε. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 231. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, νομίζω. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Είχατε δίκιο κύριε Ρικέ. Εν 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εν 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εν 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εν 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 233. ...233 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 234 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ελέγχουμε το 234. Παρακαλώ. Πέρας. Βάντεν Κάμπ. Μπράβο σας, εγκρίθηκε. Τουλάχιστον υπερψηφίσατε τη δικιά σας τροπολογία. Καλό αυτό. 236. 236 υπέρ. 236. Μα είστε άτακτοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε, δεν είναι σαφές. 249. Πέρας, απορρίπτεται. 39 απευθείας, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 253, υπέρ. Κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 255 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε τι. 255 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 255. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά εποχες εγκρινεται Εγκρίνεται. NV37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. 42 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Ένβη 39 υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά αποχές δεν ψηφίζεται πια. 263 263 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εν... NV42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 264. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV43. Δεν ψηφίζεται. 265. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβη 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, ένβη 44 έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 268 υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. 48 48 υπέρ, αποχέ, αποχές, εγκρίνεται. NV1 με συγχωρείτε, αφού εγκρίνεται πάμε απευθεία στην 51. 51, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, ψεφίζουμε την 51. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. NV2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 20-20. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία 54. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV4. NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε. NV4. Πέρας. Εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ Εξήντα πέντε, έξι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. NV6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 απευθείας. Πάνω, ε, ταυτόσιμες 78 και 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Απευθείας 6. Δεν είναι η 6, είναι η 9. NV9, υπέρ. NV9. NV9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. NV13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένβι NV14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ταυτόσιμες 15-92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 16. ένβι 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΕΝΒΙ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενενήντα επτά απευθείας. Ενενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο. Έλεγχο για την 97. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. NV19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές να ψηφίσουμε την 99. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές. Και τώρα περνάμε απευθείας στην ψηφοφορία για την διαπραγματευτική εντολή. Παρακαλώ, προσοχή. Άρχεται η ψηφοφορία για την διαπραγματευτική εντολή. Πέρας. Πέρας. «28 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, μία αποχή». Εγκρίθηκε. Κυρία Αγιούτο, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε μετά την έγκριση της δημοκρατικής εντολής. Θα σας παρακαλέσω δύο λεφτά να έχουμε ησυχία, γιατί κύριε Ντελή έχουμε πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη. Ο Υπουργός έχει φτάσει. Θέλετε να ψηφίσουμε τώρα ή να το αναβάλουμε για το απόγευμα. Θέλετε να κάνουμε τον Υπουργό να περιμένει. Ωραία. Εγώ θα κάνω ό,τι μου πείτε. Ψηφίζουμε την έκθεση του κυρίου Ντελή. Ξεκινάμε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφορία για την τροπολογία 8. Λίγη. Εγκρίνεται. Παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι σας. 110 υπέρ. Όχι καταπίπτει. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε την 115. Λίγη ψηφοφορία. Έχετε δίκιο κύριε Παντεκάπ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 150. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Λυγή εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 150. Άντε, να επαληθεύσουμε την 152. Άρχεται η σωφορία Λίγη. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Αρτού. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε το 153. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται, έχετε δίκιο. Συμβαστική 13, υπέρ. Κατά. Βοχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Όχι. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. Τροπολογία 166 υπέρ. Κατά. εποχέ Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. εποχέ Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. Επαληθεύουμε την 177. Λήξη. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. 182. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ας υπαλληθεύσουμε Την 185. Λήξη. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. εποχές. Απορρίπτεται. 187 κατά υπέρ εποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά εποχές επαληθεύουμε 188 λήξη εγκρίνεται 189 υπέρ κατά εποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 201 υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ Συγγνώμη. 204 ή 203 καταπίπτει. Ποιο είναι υπέρ τη 204 κατά εποχέ. Απορρίπτεται. 204 επαληθεύουμε λοιπόν. Λήξη. Ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 205. Υπέρ. Κατά. Συγκεντρωθείτε λιγάκι παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206 Θέλετε να επαληθεύσουμε 205. Να την επαληθεύσουμε. Κλείνω λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 209. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 2.51 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, να επαληθεύσουμε την 27. Άρχεται η συμφορία. Εγκρίνεται, έχετε και πάλι δίκιο. 28 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Ποχές. Επαληθεύουμε. Λήξη πληροφορίας. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Όχι, επαληθεύουμε την 37. Λίγη ισοφορία. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 40, 41 ξανά επαληθεύουμε. Λήξη ψηφοφορίας με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, 42 ήταν αυτή. Τώρα τη 43, υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. Σαράντα επτά υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, Αποχές. Επαληθεύουμε καλύτερα. Γιατί 48. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 δεν ψηφίζεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω τι υποτέλεσμα δίνει αυτό. Επαλήθευση. Λήξη πληροφορία για την 3. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας επαληθέψουμε. Την 82. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 84 υπέρ. Νοβότ είναι, 86 δεν ψηφίζεται. 84 υπέρ, κατά, Ποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, Ποχέ. εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, ποχέ απορρίπτεται 90 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 91 υπέρ για την 90 όχι καταπίπτουν όλες οι επόμενες περνάμε στην 93 υπέρ κατά εποχές ας υπαλληθεύσουμε Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Λήξη της 29 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Κύριε Ντελή, η έκθεσή σας εγκρίνεται. Αυτή συνάλφη. Συνεχίζουμε με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας.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 θα συζητηθεί στις μισή 17 και 30. Ε, πρόεδρε, μερικές φορές χρειάζεται για ε, λόγους ανεξαρτήτω θέλησός να πρέπει να αλλάζουμε τη μεσή διάταξη. Αλλά εγώ το απόγευμα, την ώρα που βλέπετε για τα λεωφορεία και τα πούλμαν, ε, πρέπει να βρίσκομαι στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και μου δημιουργεί πρόβλημα αυτή η αλλαγή της μεσή διάταξη. Κύριε Ντεγκράντε, Καταλαβαίνω το πρόβλημά σας. Απλά καθυστερήσαμε. Μετακινήσαμε την έκθεση Τζίλε και αν παραμείνω στο χρόνο μας θα τη διατηρήσουμε, αλλά δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Τι να σας πω. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας. Από τον κύριο Νόρμπερτ Χόφερ, Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Από την 1η Ιουλίου η Αυστρία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου με πολλές φιλοδοξίες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστριακή Προεδρία ήδη ανακοίνωσε ότι θέλει να εστιάσει την προσοχή της σε πραγματικά αυθεντικά ευρωπαϊκές λύσεις σε κοινά θέματα Εμεί εδώ σε αυτήν την επιτροπή ασχολούμαστε με θέματα καθημερινότητα των Ευρωπαϊκών πολιτών, ε, τη σύνδεση Ευρώπη. τις μεταφορές, σύνδεση των ε, περιφερειών μας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Οπότε είναι προφανές ότι η αξία της Ευρώπης αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη και για μας σε αυτή την Επιτροπή αυτή η ευρωπαϊκή αξία είναι αναμφισβήτητη. Χρειάζεται βέβαια πόρους, θέμα το οποίο θα συζητήσουμε διότι εκ παραλίλου λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό και στην Επιτροπή μας έχουμε και εμείς προτεραιότητες. Προτεραιότητα για το θέμα της ψηφιοποίησης, Γνωρίζουμε ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Δεσπόζει στην, στην επικαιρότητα. Ο τομέας των μεταφορών βρίσκεται υπό μια ταχεία μετάλλαξη εξαιτία τη ψηφιοποίηση. Γνωρίζετε ότι θα σας στηρίξουμε σε οτιδήποτε το πραγματικά ευρωπαϊκό προτείνετε και προωθήσετε. Σας δίνω το λόγο για 20 περίπου λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές για να θέσουν ερωτήματα και να τα συζητήσουμε. Μετά θα ξαναπάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Ο λόγος σε εσάς κύριε Υπουργέ, για 20 λεπτά περίπου. Σα ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι αποτελεί μεγάλη μου τιμή στο πλαίσιο της ε, σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής σας να βρίσκομαι εδώ για να σας ε, παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Αυστριακής ε, Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών και εδώ εκπροσωπώ βέβαια και την Υπουργό που είναι αρμόδια για τα ζητήματα τουρισμού και βιωσιμότητας. βέβαια έχετε μια πολύ δυναμική πρόεδρο εδώ στην Επιτροπή σας η οποία πραγματικά δείχνει μεγάλη δέσμευση για αυτά τα ζητήματα και γνωρίζει πολύ καλά τα, ότι τα όσα συζητώνται εδώ και αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ιδιαίτερη σημασία. Εμείς ε, την 1η Ιουλίου του 2018 που αναλάβαμε την ε, Προεδρία μας ω Αυστρία ε, βρεθήκαμε βέβαια σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία γιατί η διαρκή ειρήνη, η ελευθερία αλλά και η σχετική ευημερία των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ε, τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό ήταν το βασικό σκεπτικό βέβαια και των πατέρων αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή να υπάρξει μια δυναμική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζεται μια διαρκή ειρήνη και βέβαια με αυτόν τον τρόπο ε, επιτυγχάνουμε και την καλύτερη εξοικείωσή μας με την ψυχή, αν θέλετε, των άλλων εθνών της Ευρώπης, πράγμα το οποίο βέβαια καθιστά απολύτως απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των ε, διαφορετικών κρατών μελών. Και νομίζω πως αυτή είναι και η βασική προστιθέμενη, αν θέλετε, αξία της Ευρωπαϊκής Ένωση, ότι δηλαδή μπορούμε να συνεπάρχουμε παρά την πολυμορφία μας. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε μεγάλε προκλήσει, τι οποίε δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ε, κανένα κράτο μέλο ε, μόνο του. Ο διεθνή ανταγωνισμό ε, γίνεται όλο και πιο εντατικό και κατά συνέπεια ο δικό μα οικονομικό πόλο έλξη θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να διευρυνθεί. Επίσης αυξάνεται και η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και θα χρειαστεί να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα. Και βέβαια το ζήτημα της ψηφιοποίησης είναι ε, και αυτό ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει γιατί ε, και σε σχέση με αυτό τίθεται το ζήτημα ε, των πλέον εκτιμάτων των οικονομικών πόλων και της ανταγωνιστικότητας. Αν δούμε δηλαδή πώς εξελίσσεται ο κόσμος, θα δούμε πώς έχουμε από τη μία πλευρά τι ΗΠΑ, οι οποίες τώρα ε, δίνουν έμφαση στον προστατευτισμό, τη Ρωσία η οποία γίνεται ε, όλο και πιο ισχυρή και την Κίνα η οποία λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη ε, δύναμη στις διεθνείς αγορές αλλά και την Αφρική που, συχνά, που σιγά σιγά αναδεικνύεται. Άρα λοιπόν και έχουμε και την Ινδία από εκεί και μετά. Οπότε σε, στο πλαίσιο αυτού του διεθνούς ανταγωνισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ακριβώς της ενότητάς της και μέσω της ανταγωνιστικότητάς της θα πρέπει να διασφαλίσει τη δική της θέση. Και εδώ βλέπω βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κινητήρα της ε, ενοποίησης της Ευρωπαϊκής. Θα πρέπει δηλαδή και να παίρνει την πρωτοβουλία για νέες προτάσεις αλλά και να συνεχίσει το ρόλο της ως θεματοφύλακας ε, των συνθήκων. Γιατί εάν μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες θα πρέπει να πραγματικά τις ε, τηρούμε και έχουμε δει ότι με τις ε, προσπάθειες σύγκλησης ε, που κάνουμε ότι όταν υπάρχουν περίοδοι κρίσης δεν μπορούμε ακριβώς να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Οπότε αντί να αναπτύσσουμε νέα κριτήρια σύγκλησης ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να πληρούμε αυτά τα κριτήρια, γιατί ουσιαστικά τα παραβιάσαμε όλοι μας. Και νομίζω πως και το Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο Συνομοθέτης θα πρέπει να αναπτύσσουν, να δημιουργούν ε, ρεαλιστικέ λύσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν και την ευημερία αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ε, Ένωσης. Και έχω διαπιστώσει στο πλαίσιο των ε, συνομιλιών που έχουμε με Επιτροπή, με Κοινοβούλιο και με Συμβούλιο υπάρχει μια διάσταση απόψεων, δηλαδή όπου ο καθένα περιχαρακώνει τη θετική του άποψη. σω θα μπορούσαμε λοιπόν στο πλαίσιο ε, τη δική μα Προεδρία να προωθήσουμε ακριβώ μια ε, ψηλότερη, αν θέλετε, περισσότερη ενότητα ανάμεσα στου διαφορετικού εφόρου. Όπω γνωρίζετε, το σύνθημα τη Προεδρία μα είναι Ein Europa der Schutz, δηλαδή μια Ευρώπη η οποία προστατεύει. Ε, και αυτό βέβαια ισχύει και για την αύξηση της ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών. Να ε, σημειώνονται δηλαδή λιγότερα ατυχήματα. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη. Οι προσπάθειες της ε, Προεδρίας μας ε, θα στοχεύσουν δηλαδή στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περισσότερη εγκύτητα με τους πολίτες και στην περισσότερη εμπιστοσύνη από την πλευρά των πολιτών στη δυνατότητα ανάληψης δράσης της Ένωσης, αλλά και στην συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και στην εδραίωση των, ε, της σημασίας των ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Ε. Και θέλουμε εδώ βέβαια να συμβάλλουμε με, με απτό τρόπο. Και με βάση τη δική σας εμπειρία βέβαια θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι Υπουργοί ως πρόεδροι του Συμβουλίου παίζουν ένα αρκετά σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντικός είναι ο ρόλος όλου του μηχανισμού πίσω από αυτή την Προεδρία. Και εμεί έχουμε μία ε, έβρισμα λειτουργού, αν θέλετε, διοίκηση στην Αυστρία. Έχουμε δηλαδή εδώ μία σειρά από συνεργάτε μα, οι οποίοι συνεργάζονται, οι οποίοι συμμετέχουν σε όλε τι συνεδριάσει, προκειμένου να επιτυχάνουμε συμβιβασμού, προκειμένου να φτάσουμε σε μία συμφωνία. Άρα λοιπόν εδώ εμπιστεύομαι όλο το προσωπικό τη διοίκηση μα γιατί εκείνοι είναι εκείνοι οι οποίοι διασφαλίζουν τελικά την, ε, την επίτευξη μιας συμφωνίας. Δεν είναι οι υπουργοί οι οποίοι φτάνουν στη συμφωνία. Εκείνοι είναι, αν θέλετε, που υπογράφουν τη συμφωνία, αλλά εκείνοι που την επιτυχάνουν στην πραγματικότητα στα παρασκήνια είναι ε, εκείνοι που δεν φαίνονται και συχνά στα πόδια της δημοσιότητας. Ε, τώρα, θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι βασικέ προτεραιότητε μα στον χώρο των μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε περισσότερο τα αισθήματα μεταφορών προκειμένου να έχουμε έναν δίκαιο και ισορροπημένο ανταγωνισμό. Θέλουμε ταυτόχρονα ε, ένα δίκαιο και υψηλό επίπεδο ε, συνθήκων εργασίας αλλά και κοινωνικών συνθήκων. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε περαιτέρω την ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών και θέλουμε να συμβάλλουμε από την πλευρά μα στην πιο βιώσιμη κινητικότητα που θα λαμβάνει υπόψη και την κλιματική μεταβολή. Ε, εμείς θεωρούμε λοιπόν τη δική μας ε, Προεδρία ως μια Προεδρία εργασία των εισαγωγικών. Δηλαδή ε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί των νομοθετικών προτάσεων που γίνονται. Ωστόσο, φυσικά θα δώσουμε προτεραιότητα στις προτάσεις εκείνες όπου μπορούμε να επιτύχουμε ρεαλιστική πρόοδο. Και φυσικά ο τακτικός και ανοιχτός διάλογος με το Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή αποτελεί το, τη βασική προϋπόθεση για να φτάσουμε σε πρακτικές λύσεις έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μιας ε, ε, σύγχρονης, μιας ε, σύγχρονης οικονομίας αλλά και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση βέβαια στη βελτίωση των κοινωνικών και οικολογικών παραμέτρων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την ε, προηγούμενη, τη Βουλγαρική Προεδρία για τα όσα έκανε προκειμένου να προωθήσει ε, τις ε, νομοθετικές προτάσεις που συζητούμε αυτή την περίοδο. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το οποίο τώρα αναλαμβάνουμε εμείς να κάνουμε και πραγματικά ευχαριστώ θερμά τη Βουλγαρική Προεδρία για όσα έκανε μέχρι τώρα. Εμείς από την πλευρά της Αυστρίας ε, έχουμε αναλάβει και στο παρελθόν την Προεδρία του Συμβουλίου, είναι τρίτη Προεδρία που αναλαμβάνουμε ε, και ε, το Κοινοβούλιο ασχολείται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις χειρισίες μεταφορές με τα πακέτα κινητικότητας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρώτο πακέτο κινητικότητας αναλύσαμε ακριβώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση στην εργασία και στην ε, αγορά μεταφορών σε ό,τι αφορά τους χρόνους ανάπαυσης και τους χρόνους οδήγησης, τους ε, ταχογράφους, την επιβολή των κοινωνικών διατάξεων, αλλά και το Lex Specialis. Επίσης, αναλύουμε πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα σημεία αυτών των προτάσεων, έτσι ώστε να δούμε πού διαγράφονται, πού διαφαίνονται ρεαλιστικοί συμβιβασμοί έτσι ώστε τελικά να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες ε, ε, πλειοψηφίε για την επίτευξη ε, ενός συμβιβασμού. Πραγματικά σας λέω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε εδώ σε βιώσιμους συμβιβασμούς. Και σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σε εντατικό διάλογο και σε διμερείς επαφές με όλους τους stakeholders, όλους τους συναμόδιους φορείς και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση εδώ στις τοποθετήσεις του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τους επιμέρους φακέλους ακόμα και αν δεν βρισκόμαστε ακόμα βέβαια στη φάση των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή για μας είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε τις εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αντιλαμβανόμαστε τα κίνητρα για τι τοποθετήσει αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς με σφαιρικό τρόπο το status quo του, πού βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι για να φτάσουμε ε, σε επιτυχίες της περαιτέρω, στις περαιτέρω συζητήσεις. Και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, επαναπροωθήθηκε, ουσιαστικά απορρίπτηκε από την Ολομέλεια η σχετική ε, ε, πρόταση στην Επιτροπή Τραν, καταδεικνύει το πόσο περίπλοκος είναι αυτός ο τομέας και πόσο απαραίτητο είναι να βρούμε εδώ τις σωστές προτάσεις. Άρα λοιπόν εμείς από την πλευρά της Προεδρίας μας θα εργαστούμε με συνέπεια και θα προσπαθήσουμε στο πλαίσιο ε, του Συμβουλίου Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Ενέργεια ε, του Δεκεμβρίου να φτάσουμε σε ένα γενικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά αυτού του φακέλου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμεί από την πλευρά τη Αυστρία, ε, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια καλή λύση και να και βέβαια γνωρίζετε ότι ο τριμερής διάλογος με το Κοινοβούλιο ξεκινάει αύριο στις 11 Ιουλίου και θεωρώ πω εδώ υπάρχουν καλές προοπτικέ για να φτάσουμε σε επιτυχία εκβασή των διαπραγματεύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα άλλο φάκελο του πρώτου ε, πακέτου ε, κινητικότητας, ε, δυστυχώς οι απόψει και μεταξύ των διαφορετικών κρατομελών είναι πιο ε, ε, δηλαδή, το κατά πόσο θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας, το Eurovinet δηλαδή, να καλύπτει και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ε, με βάση δηλαδή τα όσα λαμβάνουν υπόψη τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη διατήρηση εδώ της επικουρικότητας και σε σχέση με αυτές τις προτάσεις ε, που γίνονται, ε, θεωρείται λοιπόν αυτό το ζήτημα προβληματικό από πολλά κράτη-μέλη. Και γνωρίζετε βέβαια και την άποψη της Αυστρίας σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, στο πλαίσιο εμείς της Προεδρίας που αναλαμβάνουμε, θέλουμε να είμαστε ένας αμερόληπτος διαμεσολαβητής και όχι να προωθήσουμε τη δική μας ε, άποψη ως κράτος μέλος. Και αυτό πραγματικά σας το υπόσχομαι με ειλικρίνεια. Ε, λόγω των διαφορετικών απόψεων, που υπάρχουν και αρκετά διστάμενων απόψεων, ε, δεν νομίζω πως θα είναι εύκολο να επιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά πάντα την Ευρωβινιέτα. Ε, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την της, τον κοινωνικό πυλώνα και τον πυλώνα σε ό,τι αφορά την ε, αγορά αυτού του ε, πακέτου θα ε, έρθω σε περισσότερες λεπτομέρειες τώρα στα επόμενα πακέτα κινητικότητα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πακέτο κινητικότητα, έχουμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο βέβαια επεξεργάστηκε εντατικά η Βουλγαρική Προεδρία, δηλαδή την πρόταση για μια νέα πρόταση σε ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές. Από ό,τι γνωρίζω αυτή η πρόταση είναι πολύ σημαντική και για σας, για την Επιτροπή σας και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών τρόπων μεταφορών και βέβαια γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν και σχετικές ε, διαπραγματεύσεις εντός ε, του ε, Κοινοβουλίου και νομίζω πως και η δική σας Επιτροπή έχει διαβουλευτεί λεπτομερώς από αυτού του ζητήματος. Εμείς λοιπόν από τη δική μας πλευρά παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις τοποθετήσεις του Κοινοβουλίου και το, στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θέλουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία έτσι ώστε να ξεκινήσουν ταχύτατα διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο ε, και προκειμένου να ολοκληρωθούν ή δυνατόν ε, υπό τη Ρουμανική Προεδρία. Ένα, ένας περαιτέρω τώρα φάκελος, επί το οποίο ψηφίσατε νομίζω σήμερα το πρωί, στην Επιτροπή σας και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ε, ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών είναι βέβαια το ζήτημα ε, της οδηγίας για τα καθαρά αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο δηλαδή ε, των στόχων που έχουμε θέσει για την προώθηση των αυτοκινήτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές και την τι περαιτέρω αγορέ τέτοιων οχημάτων και στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, εμεί από την πλευρά μα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο σε σχέση με αυτό το φάκελο αλλά επειδή η συζήτηση στο επίπεδο του Συμβουλίου βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, δεν πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε πραγματικά σε μια συμφωνία στο πλαίσιο τη δική μα Προεδρία, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τρίτο τμήμα ε, του πακέτου κινητικότητα, ε, ε, θα δώσουμε προτεραιότητα στις προτάσει ό,τι αφορά την αύξηση τη ε, ασφάλεια ε, στι ε, μεταφορέ, προκειμένου βέβαια να λάβουμε υπόψη μα και τι πρόσφατε εξελίξει σε ό,τι αφορά το, την αυτομετωπιμένη και την διαδικτυωμένη οδήγηση. Εδώ μιλάμε δηλαδή για την αναθεώρηση τη γενική οδηγία ασφαλείας και την οδηγία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τη υποδομή. Οι διαπραγματεύσει στις σχετικέ ομάδες εργασία του Συμβουλίου έχουν ξεκινήσει και η, ο στόχο τη προεδρία μα είναι να φτάσουμε σε ένα, γενικό, μια γενική, ένα γενικό προσανατολισμό από την πλευρά του Συμβουλίου. Καθώ ε, λοιπόν μια αποτελεσματική υποδομή αποτελεί προπόθεση για ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό σύστημα κινητικότητα, ε, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στι ε, διατάξει που αφορούν το χώρο των μεταφορών του κανονισμού για το ΣΕΦ, για το χρηματοδοτικό δηλαδή μηχανισμό συνότητα Ευρώπη και ε, την πρόταση σε ό,τι αφορά την ε, προώθηση τη εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορά. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να διασφαλιστεί και κατάλληλη χρηματοδοτική πρικοδότηση τη δεύτερη γενιά του ΣΕΦ και θα πρέπει και οι δυνητικέ ε, συγχρηματοδοτήσει να διασφαλιστούν σε ό,τι αφορά και την περαιτέρω προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών τρόπων μεταφορά αλλά και προκειμένου να ληφθούν υπόψη και οι απόκεντρε περιοχέ καθώς πρόκειται εδώ για ένα σημαντικό εργαλείο για ε, μια ε, πολιτική μεταφορών και υποδομής η οποία είναι και βιώσιμη αλλά λαμβάνει υπόψη της και τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα. Στον τομέα βέβαια της ε, αεροπορίας, στον οποίο και εγώ, από τον οποίο προέρχομαι αν θέλετε πανδηματικά, εδώ θέλουμε να επιτύχουμε μια σημαντική πρόοδο προκειμένου να ενισχύσουμε την Ευρώπη ω οικονομικό πόλο έλεξη και θα ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αεροπορία. Ε, πρόσφατα στι 7 Ιουνίου το Συμβούλιο, οι Υπουργοί δηλαδή Μεταφορών έφτασαν σε μια συμφωνία ε, και εμεί θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια λοιπόν αυτή τη συμφωνία να φτάσουμε σε μια βιώσιμη ε, λύση που θα αποβεί προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής οικονομίας και των εργαζομένων μας. Και η Αυστριακή Προεδρία θα παρακολουθήσει βέβαια και πολύ προσεκτικά την εντολή της Επιτροπής ε, και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για γενικές ε, συμφωνίες ε, αναίρεσης κυκλοφορίας με τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ναυσιβλοίας, προφανώς εμείς δεν έχουμε κάποια ε, άμεση εμπλοκή εδώ, αλλά στο πλαίσιο τη δική μα προεδρία θα εστιάσουμε και στον, ε, στην αυσιπλοεία στις εσωτερικέ οδούς ε, και στην ε, θαλάσσια αυσιπλοεία. Θέλουμε να υπάρξουν εδώ συμπεράσματα του Συμβουλίου, ε, προκειμένου η συμβολή της αυσιπλοείας στις εσωτερικέ πλωτές οδούς στις ε, πολυτροπικές μεταφορές να αυξηθεί. Και ε, στον τομέα της, ε, των θαλάσσιων, θαλάσσιας πλοίας θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση σε ό,τι αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής έτσι ώστε στα τέλη του έτους να φτάσουμε σε συμφωνία. Επίσης θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα γενικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά την πρόταση για ένα κανονισμό για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου single window έτσι ώστε να επιτύχουμε και σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά και την ε, οδηγία για την ε, αλλαγή των υφιστάμενων οδηγιών σε ό,τι αφορά τι ελάχιστε απαιτήσει κατάρτιση των ναυτικών και την αμοιβή αναγνώριση των πιστοποιητικών του. Και επίση στο σχετικό συμβούλιο των Υπουργών στι 3 ε, Δεκεμβρίου στι Βρυξέλλε ε, θα γίνει σχετική συζήτηση. Στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, ή μάλλον παράλληλα με αυτό, θα λάβει η χώρα και η συνεδρίαση των κρατών από τα οποία διέρχεται ο ε, Δούναβη. Και επίση να σα ενημερώσω ότι στι 29 και 30 Οκτωβρίου του 2018 στο Γκράτ θα λάβει η χώρα ένα άτυπο Υποσυμβούλιο Υπουργών ε, Μεταφορών και ε, Περιβάλλοντος ε, που θα εστιάσει στα κύρια θεματικά πεδία μείωση των ατρακούχων εκπομπών, ασφάλεια των μεταφορών, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πολυτροπικότητα των μεταφορών. Άρα λοιπόν ε, το τα, ζητήματα που θα καλύψουν καλύπτουν ένα ευρύ ε, φάσμα περνώντα από τις, από τις γενικότερες μεταφορές σε ό,τι αφορά την προστασία του κλίματος, ε, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας και φτάνοντας ως τον τομέα της υποδομής. Και βέβαια θα υπάρξει και αυτή, όπως είπα, η άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών διατομεακά έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε, να βάλουμε και το δικό μας πετραδάκι αν θέλετε σε αυτή τη γενικότερη προσπάθεια και ενδεχομένως να αποτελέσει και ορόσημο αυτή η Προεδρία μας για την πρόοδο που θα επιτύχουμε ε, σε ό,τι αφορά ένα ε, βιώσιμο σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Ε, Ολοκληρώνοντα την παρουσίαση που κάνω σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, θα ήθελα να σα πω πόσο σημαντικέ θεωρούμε τι επαφέ μα με το Κοινοβούλιο από την πλευρά τη Αυστριακή Προεδρία. Και θα ήθελα να σα πω εδώ ότι υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό στόχο από την δική μα πλευρά. Θέλουμε λοιπόν με την Προεδρία μα και στο πλαίσιο του παραδοσιακού ρόλου που αναλαμβάνουμε να δράσουμε ω διαμεσολαβητή ω γεφυροποιός εντό εισαγωγικών προκειμένου να ε, συμβάλλουμε και εμεί στην περαιτέρω ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα επιτρέψτε μου κυρίε και κύριοι εκπροσωπώντα ε, την αξιότιμη συνάδελφό μου, την ε, Ομοσπονδιακή δηλαδή Υπουργό Ελίζαμπεθ Κιώστιγκερ, η οποία λόγω τη γέννηση του πρώτου σου παιδιού δεν ε, μπορούσε να παραβρίσκεται εδώ, να σα κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τον ε, τομέα του τουρισμού και ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, και καταρχήν θα ήθελα να σα ε, μεταφέρω ε, του θερμούς χαιρετισμούς τη συναδέλφου του Υπουργού, η οποία βέβαια διατέλεσε και ω Ευρωβουλευτή, κατά συνέπεια γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία αυτού του φορέα. Οι τρέχουσες λοιπόν εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού καταδεικνύουν ότι ο τουρισμός στις περισσότερες περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την οικονομία. Δηλαδή δημιουργεί προστιθέμενη αξία, αλλά και ειδικότερα στι περιοχές, αλλά και θέσει δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού. Ε, και επίση συνδέει του ανθρώπου ε, και προωθεί την πολιτισμική ανταλλαγή. Ε, σε κατά κύριο λόγο βέβαια αποτελεί εδώ ο τουρισμός ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών, των περιφερειών και των ε, τοπικών αρχών, πράγμα το οποίο είναι καλό λαμβάνοντα υπόψη ε, την επικουρικότητα. Αλλά υπάρχουν στοιχεία όπως η εσωτερική αγορά, η καινοτομία, η περιφερειακή ανάπτυξη, η απέντηση στους ανθρώπους, η εκπαίδευση, η πολιτισμική και η φυσική πόρη, το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ζητήματα τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουν βέβαια ιδιαίτερη σημασία για να βιώσιμο αλλά και ανταγωνιστικό ε, τουρισμό. Και κατά συνέπεια θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στον τουρισμό. Ε, λόγω του, του μεγέθους του ε, αλλά και της δυναμική του ανάπτυξη, αυτό ο τομέας θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης και να είναι προσαρμοσμένα στι ανάγκες του αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρω το δυναμικό του. Και βέβαια, α μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη μέσα τάξη στην Κίνα, στην Ινδία, ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι έχουν πλέον περισσότερο χρόνο και δυνατότητε να ταξιδέψουν. Άρα λοιπόν ο τουρισμό έχει μεγάλη σημασία και για το μέλλον. Θα πρέπει ε, να έχουμε βέβαια ταυτόχρονα πάντοτε υπόψη μα τι συνθήκε που θα επικρατούν για τα 2 εκατομμύρια ε, πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Και βέβαια εμεί δίνουμε ιδιαίτερο, ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το μέγεθο επιχειρήσεων. Δηλαδή το νέο πλαίσιο δεν θα πρέπει να προβλέπει ε, περιτέ και πολύ επαχθείς ε, διατάξεις για αυτέ τι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Στο πλαίσιο λοιπόν τη Προεδρία μα θα εστιάσουμε στην επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων εφορέων και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσουμε στα, στις αρχές του Οκτωβρίου το 17ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού στη Βιέννη όπου θα συζητήσουμε ποιες είναι οι στρατηγικές για τον τουρισμό που μπορούμε να αναπτύξουμε έτσι ώστε να ε, αυξήσουμε μακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής αλλά και την παραγωγή προσθέμενης αξίας και βέβαια είστε θερμά προσκεκλημένοι σε αυτό το ε, φόρουμ. Ζητώ συγγνώμη, ε, κύριε Πρόεδρε, άμα λίγο. Και θα ήθελα εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσω για την, ε, είμαι βέβαιος, επικοδομητική συνεργασία που θα έχουμε κατά τους επόμενους μήνες ε, και είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε πάρα, πολλά από κοινού και ε, είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε Υπουργέ. Χρησιμοποιήσατε κουβέντε που καλό είναι να τι κρατήσουμε. Μιλήσατε για προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, μιλήσατε για τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού μέλλοντος, για την ειρήνη στην Ευρώπη. Θυμήσατε ότι χρειάζεται μια Ευρώπη που προστατεύει. Είπατε ότι είναι πια καιρό να υλοποιηθούν νέε πρωτοβουλίε σύγκληση. Ωραίο ενθουσιασμό εκφράσατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να είναι επικοδομητικό. διότι οι προκλήσει, όπω είπατε, είναι σοβαρέ. Ιδίω, όπως είπατε, το πακέτο για την κινητικότητα, όπου άκουσα να χρησιμοποιείτε τον όρο, θα μας το εξηγήσετε και στο Συμβούλιο, είπατε ότι θα κάνετε προτάσεις, κυρίως προτάσεις συνδυαστικές. Το ερώτημα είναι πώς θα φτάσουμε, έστω και με σήματα καπνού, να έχουμε μια συμφωνία για την ε, ε, κινητικότητα στο Συμβούλιο και είπατε ότι και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι κάτι που θα φανεί με την προηγμένη διασύνδεση των ευρωπαϊκών κρατών. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση με πρώτο τον συνάδελφό μας τον κύριο Βάντεν Κάμπ. Κύριε Κάμπ, να σας το πω, όπως θα το πω και σε όλους τους ε, συναδέλφους, ο χρόνος σας είναι περιορισμένος στα δύο λεπτά. Ναι, ναι, δύο λεπτά. Γιατί θέλουν κι άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Οι οποίοι θα έχουν το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Βαντενκάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ΕΛΚ καλωσορίζει την Αυστριακή Προεδρία και τον Υπουργό κ. Χόφερ, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γνωρίζουμε ότι η Αυστρία αυτή τη στιγμή έχει κυβέρνηση συνασπισμού, ετερόκλητου συμβασμού και γνωρίζω ότι αυτό είναι επικίνδυνο για αυτό που αναλαμβάνεται. Εξετάζοντα τι εξελίξει τη ΗΠΑ, στην Κίνα, την Ινδία, ε, για αυτές τις χώρες είμαστε ο αδύναμος εταίρος. Χρειαζόμαστε λοιπόν η Αυστρία να δομήσει τις σχέσεις μας με τρόπο ώστε να ενισχύσουμε τη θέση μα, Το πακέτο θα πρέπει να είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι γνωστή η θέση τη Αυστρίας για τα διόδια, για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Καλή επιτυχία. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι είπατε για το συνέοντα στην Ευρώπη. Ο κ. Κόρτ, ο καγκελάριο σα, ε, ζητάει περικοπέ. Πώς θα γίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά τις ε, ποτάμιες οδούς, ελπίζω ότι μπορούμε να τις αναπτύξουμε μέσω του Δούναβη σε ε, μεγαλύτερο βαθμό. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κώστιγκερ. Επίσης, ο τουρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Αυστρία. Αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε καινούρια εμπόδια στην κινητικότητα ε, των οχημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρασφάλα Χάνης τώρα. Σας ευχαριστώ ε, και σας καλωσορίζουμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ε, εξέτασα το πρόγραμμα της Προεδρίας σας και νομίζω πως είναι αρκετά μετριοπαθές αν θέλετε, δηλαδή μόνο μία σελίδα αφορά τις μεταφορές και είναι γενική αυτή η στόχη και όχι συγκεκριμένη. Πάντως ένας από αυτούς που αναφέρεται είναι οι συνθήκες εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες. Έχουμε δει όμως πώς ψηφίζουν τα ε, ε, Πολιτικέ ομάδε, ε, δηλαδή και συγκεκριμένα το FAOP και το FP, ε, ε, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω πω διαφοροποιούνται οι απόψεις του από αυτό που θέλετε να προωθήσετε εδώ στην Προεδρία. Ειδικότερα, για παράδειγμα, η περισσότερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την περιόδου ανάπαυσης και εργασία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, στο οποίο θα πρέπει να αντιταχθούμε. Ωστόσο, μια σχετική απόφαση λήφθη από το Συμβούλιο εδώ, παρότι υπήρξαν μαζικέ αντιστάσει και χωρί να ληφθούν υπόψη οι συλλογικοί εταίροι συγκεκριμένα ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω. Άρα λοιπόν, οι διαφορετικές, διαφορετικοί τοποθετήσει σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μεταφορών από τα πολιτικά κόμματα FAP, ε, FPE, ε, ε, ε, καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή από τη δική σα πλευρά. Οπότε θα ήθελα να γνωρίζω από τη δική σα πλευρά ε, ποια είναι η δική σα θέση σε ό,τι αφορά αυτά στου σημαντικού φακέλου, απόσπαση δηλαδή οδηγών και χρόνοι ανάπαυσης και εργασίας. Έχετε εδώ μία κοινή γραμμή ή τι ακριβώ θέλετε να επιτύχετε. Ε, θέλετε να εξαιρέσετε τελείω ε, ε, τι διεθνεί μεταφορές ή τι ακριβώ θέλετε να προβλέψετε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αποσπάσει των εργαζομένων. Ένα ακόμα ερώτημα τώρα. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θέλετε να λάβετε στο πλαίσιο τη Προεδρία σας σε ό,τι αφορά ε, το κοινωνικό dumping στους, ε, στις οδικές αρτηρίες της Ευρώπης. Και επίσης ένα ακόμα ε, σε ό,τι αφορά την, το ανώτατο όριο των 12 ωρών εργασίας ανά ημέρα. Υπάρχει κάτι τέτοιο, μια πρόβλεψη σε ό,τι αφορά του επαγγελματικού οδηγού ε, στην Ευρώπη και επίση σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασία. Εσεί θα ήσασταν διατεθειμένο ε, να ε, συμφωνήσετε με την εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων προκειμένου αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να μπορέσει να αναλάβει δράση κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ένα ακόμα ερώτημα θα ήθελα να θέσω σε ό,τι αφορά ε, την Βρένα και το ε, ζήτημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί στο, στο πληθυσμό να υποφέρει. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θέλετε να λάβετε ως ε, Υπουργό προκειμένου το, όλο αυτό το πρόβλημα του τράντζι στο Βρένα να μειωθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από λίγες εβδομάδες πήγαμε στη Βιέννη σε μια διάσκεψη του Προεδρείου και συζητήσαμε και το βασικό θέμα της Προεδρίας σας, Ευρώπη που προστατεύει. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες κατάστασεις, ε, καταστάσεις ρεψοκίνδυνες σε σχέση με την κινητικότητα. Το ερώτημα είναι πώς προστατεύουμε και πόσο μπορούμε να προωθήσουμε την κινητικότητα. Όπως ξέρετε, οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές είναι υπέρ της ενιαίας αγοράς. Ε, γι' αυτό μας απασχολούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις εδώ στο Κοινοβούλιο για τέτοια θέματα διότι είναι μια πολύ λεπτή γραμμή αυτή η διαχωριστική γραμμή για τη νέα νομοθεσία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές προποθέσει, αλλά και την προστασία της ενιαίας αγοράς που δεν πρέπει να γίνεται προστατευτισμός. Γι' αυτό λοιπόν η θέση σας στο πακέτο περί κινητικότητας ε, δεν ε, πέρασε ακριβώ. Αν και ε, είχαμε μια καλή συμβαστική ω Επιτροπή Μεταφορών για το πακέτο κινητικότητα στην Ολομέλεια, χάσαμε. Και ω Προεδρία του Συμβουλίου, όπω περιγράψατε ε, τον εαυτό σα θα είσαστε μια ε, εξελίξη εργαζόμενη Προεδρία, θα πρέπει να δούμε πόσο θα μπορείτε να διαπραγματευτείτε, γιατί επίκενται και εκλογέ μετά το διάστημα τη δική σα Προεδρία. Τέλο πάντων, για το πακέτο τη κινητικότητα όπω το περιγράψατε, λέτε ότι πήρατε τα στοιχεία τη Βουλγαρική Προεδρία για, να προχωρήσετε, για να προχωρήσετε στο δεύτερο πακέτο. Ε, στο δεύτερο πακέτο κινητικότητας και την ε, πρόσβαση στην αγορά που είναι η δική μου έκθεση, τι σκοπεύετε να διοργανώσετε για το θέμα αυτό. Διότι θα θέλαμε να προλάβουμε μέσα σε αυτή τη θητεία το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την ε, τοποθέτηση του σε πρώτη αναγνώση για την ε, διευκόλυνση τη σύνδεση τη Ευρώπη. Είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κονδύλια και είναι σημαντικό για το δίκτυο μεταφορών, αλλά πρέπει να ξοδευτούν σε συνδυασμό με τα, με τα κονδύλια τη συνοχή. Μας ενδιαφέρει εδώ η αντίδρασή σας και σε σχέση με τη στρατιωτική κινητικότητα. η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και τα λοιπά λέτε ότι αυξάνουν τον προπολογισμό του. Στη Ρωσία δεν ισχύει αυτό μόνο σε ένα τομέα. Τα στρατητικά ε, εκεί ε, δίνουν περισσότερα οι Ρώσοι. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε και στην Ευρώπη. Ε, Σα ευχαριστούμε κύριε Ζήλε. Παρότι μιλήσατε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε, ο κύριο Τέλη έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ και σας χαιρετίζω και από την πλευρά της Άλντε. Ε, θα ήθελα να πω ότι έχουμε την αίσθηση ότι η, Αυστρία, η Αυστριακή Προεδρία δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον ε, προκειμένου να επιτευχθεί μια πρόοδο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και πραγματικά έχετε αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορείτε να δράσετε ως διαμεσολαβητής. Το αναφέρατε κι εσείς ε, κατά την έναξη της ομιλίας σας και θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που ανέφερε ο κύριος Ζήλερ. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δευτερεύον σύνθημα, θέλετε, από την πλευρά τη ε, Πρόεδρε, δηλαδή σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θέλουμε βέβαια να δώσουμε το λανθασμένο μήνυμα ότι είμαστε υπερβολικοί εδώ. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε πραγματικά είναι περισσότερη ανταγωνιστικότητα και η τη οικονομική ισχύω τη Ευρώπη και νομίζω πω και την αξιοποίηση του οικονομικού του δυναμικού. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να πούμε τώρα. Αναφερθήκατε στι προτεραιότητε που θέλετε να δώσετε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά φακέλου όπου μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο. Ε, Όμω θα ήθελα να πω και το είπατε και ρητά, ότι σε σχέση με το πακέτο κινητικότητας ε, θέλετε να ε, πετύχετε πρόοδο και θα πρέπει να υπάρξει και μια έκθεση πρόοδου σε ό,τι αφορά ε, παρότι βέβαια το ότι αναφέρθηκε εδώ κάτι για την προηγούμενη εβδομάδα ενδεχομένω να δημιουργεί λαθασμένε εντυπώσει. Πάντω, σε ό,τι αφορά την πρόοδο σε σχέση με ε, του δύο σχετικού φακέλου στου οποίου αναφερθήκατε, εδώ ε, δεν ξέρουμε ακριβώ αν μπορούμε να κρίνουμε από το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Δηλαδή, καταρχήν θα πρέπει να δούμε ειδικότερα σε ό,τι αφορά του ε, αποσπασμένου εργαζόμενου το τι χρειάζεται εδώ να ε, διορθώσουμε. Και εδώ τίθεται και το ζήτημα του. Ε, ότι δηλαδή από τη μία πλευρά σε ό,τι αφορά το καμποτάζ η κατάσταση είναι τελείω διαφορετική σε ό,τι αφορά τη συνένεση από ό,τι σε ό,τι αφορά την πρόταση για του αποσπασμένου εργαζομένου. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα τελευταίο ερώτημα, μπορούμε να εστιάσουμε ε, τι συμβαστικές τροπολογίες ε, οι οποίε έχουν τεθεί και στο πλαίσιο τη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου γιατί ε, αυτέ οι συμβαστικέ τροπολογίες είναι ουσιαστικά εκείνες που περιέχουν τι βασικέ γραμμέ τη σκέψη του Κοινοβουλίου και αν μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτέ, νομίζω πω θα υπάρξει περαιτέρω ενθάρρυνση για την επίτευξη πρόοδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τέλητσκα για αυτά τα ερωτήματα. Δίνω το λόγο στον κύριο Κράμερ. Σα ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ε, παρουσίαση. Αναφερθήκατε στη μείωση των ανθρακών εκπομπών από το τομέα ε, των μεταφορών και αυτό είναι σημαντικό για μα. Αναφερθήκατε και στα διόδια εδώ ε, και φυσικά εδώ υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσει από την πλευρά των κρατών μελών. Οπότε ελπίζω ε, η Αυστρία να υποστηρίξει την προσφυγή που έχει γίνει σε ό,τι αφορά αυτή την επιβολή των διοδίων σε, σε αλλοδαπούς. δηλαδή, ε, ουσιαστικά ε, είναι ε, σκανδαλώδες το γεγονός ότι για κάθε ξεχωριστό χιλιόμετρο σιδηροδρόμου έχουμε την επιβολή τέλους ε, διοδίων ενώ σε ό,τι αφορά τους αυτοκινητοδρόμους μόνο το 1% για το 1% είσαι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι ουσιαστικά ε, υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά διάφορες λύσεις οι οποίες δεν είναι φιλοπεριβαλλοντικές ενώ τις φιλοπεριβαλλοντικές δεν τις υποστηρίζουμε. Τώρα, ε, από εκεί και μετά έχουμε σε ό,τι αφορά τα φορτηγά έχουμε μία σειρά από επιχειρήσει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ε, παράδοση δεμάτων, οι οποίε έχουν ε, μετατρέψει αντίστοιχα ε, τα, τα φορτηγά του. Και νομίζω πω θα πρέπει να ισχύσει μία γενικότερη υποχρέωση, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τα ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα. Ε, τώρα, ένα ακόμα ζήτημα. Η χρηματοδότηση μέσω ΣΕΦ. Νομίζω ε, πω η χρηματοδότηση είναι επαρκή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 30 χρόνια. Ε, ε, επενδύουμε ε, πάρα πολλά στο να είμαστε ενωμένοι ως Ευρώπη, αλλά υπάρχουν πάρα πάρα πολλά κενά στο συνδρομικό δίκτυο. Ε, και βέβαια ε, έχετε είναι δύσκολο για σας να πείτε στα υπόλοιπα κράτη-μέλη να κλείσουν αυτά τα κενά που έχουν στο δικό του συνδρομικό δίκτυο, γιατί δεν το κάνετε εσεί ήδη ως ω Αυστρία. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά και σύνδεση, για παράδειγμα, βγαίνει Πράγα. Δηλαδή, μετά από την, την, την μετά από το σιδηρούν παραπέτασμα ουσιαστικά δεν έχει γίνει καμία πρόοδο εκεί προκειμένου να κλείσει αυτό το κενό. Οπότε σα ρωτάω ευθέω ω Υπουργό Μεταφορών, θα ήσασταν διατεθειμένο να ε, ξεκινήσει και πάλι αυτή η σύνδεση, έτσι ώστε να δώσετε το καλό παράδειγμα και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρώπη. Ε, τώρα, δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα του πακέτου κινητικότητα, αλλά υπάρχει μία βασική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίδιο επίπεδο μισθού για την ίδια εργασία στο ίδιο σημείο εργασία. Ε, εντάξει, αυτό μπορεί να μην ισχύει για όλου του οδηγού ε, φορτηγών, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύει ω αρχή. Δηλαδή, εάν μια νοσοκόμα ε, που προέρχεται από τη Ρουμανία ε, εργάζεται στη Βιέννη, δεν θα τη πείτε όχι, είστε από τη Ρουμανία, άρα θα σα πληρώσουμε τα μισά. Η ίδια λογική λοιπόν θα πρέπει να ισχύει και για του οδηγού ε, των φορτηγών και των επαγγελματικών. Οπότε θα ήθελα να ακούσω ποια είναι δική σα θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ, τον κύριο Σμάια. Ευχαριστώ. Ε, Δυστυχώ έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για τι παρεμβάσει μα. Ε, καταρχήν, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά, κύριε Υπουργέ, εδώ στην Επιτροπή μα, ε, αλλά και στο Κοινοβούλιο. Ε, γενικότερα, γνωρίζω ότι ε, θα συναντήσετε και άλλου συναδέλφου σήμερα εδώ. Οπότε. Ε, Ευχαριστούμε ε, για το γεγονό ότι ε, δίνετε ιδιαίτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Μα είπατε ήδη ότι ε, είχατε, αναλαμβάνετε για τρίτη φορά την Προεδρία της, του Συμβουλίου και βέβαια σε δύο από αυτέ τι προεδρίε εγώ είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα μας είπατε σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών και βέβαια ε, έχουμε μια κάπως διαφορετική ε, προσέγγιση ό,τι αφορά τα διάφορα ζητήματα, αλλά εκείνο που θεωρώ λυπηρό είναι το γεγονός ότι η ε, σοσιαλιστική ομάδα ουσιαστικά έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από το κοινό πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Και βέβαια εμείς απορρίψαμε αυτό το πακέτο την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπατε και εσείς στην Ολομέλεια, γιατί θεωρήσαμε ότι ε, ορισμένα συζητήματα σε ό,τι αφορά τις κοινωνικέ συνθήκε είναι απαράδεκτα. Πάντως, ε, ε, μας είπατε ότι το σύνθημα της Προεδρίας σας είναι μια Ευρώπη η οποία προστατεύει. Πώς λοιπόν θα εκφραστεί αυτό το σύνθημά σα αυτή η αρχή στην πολιτική μεταφορών από εκεί και μετά, εσεί θεωρείστε ω Αυστρία ένα κράτο μέλο το οποίο αναλαμβάνει ιδιαίτερη δράση στον τομέα των μεταφορών. Πώ λοιπόν θεωρείτε πω μπορούμε να αυξήσουμε την ασφάλεια στου στους, ε, ε, δρόμου τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχουμε λιγότερα ατυχήματα και λιγότερα δυστυχήματα και θανάτου. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω ε, πώ βλέπετε τι περαιτέρω εξελίξει και μελλοντικέ εξελίξει στον τομέα τη αυτοματοποιημένη και διαδικτυωμένη οδήγηση. Θα θέσετε συγκεκριμένε προτεραιότητε στη ε, δική σα ε, Προεδρία, γιατί βέβαια ε, μέσα στο 2017 έτρεξε στη δική μου πόλη, στο Κράτ, ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα. Ένα τέταρτο ερώτημα είναι το εξή. Σε ό,τι αφορά την μεταβίβαση των εμπορευματικών μεταφορών από τι οδικέ μεταφορέ στι ιδρωμικέ μεταφορέ, εδώ ήδη έχουμε αναλάβει ηγετικό ρόλο. Είμαστε στο 32% για παράδειγμα, ενώ ε, το μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 20%. Τι μπορούμε λοιπόν να δείξουμε ε, σε ό,τι αφορά αυτήν την ε, μεταβίβαση και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην διατύπωση της οδηγίας για τις συντηρησμένες μεταφορές. Ευχαριστώ, λέω ο Πρόεδρο. Είμαστε ακόμα στου συντονιστέ. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Γιούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, Υπουργέ. να σας πω ότι είμαι εισηγήτρια για τις συνδυασμένε μεταφορές και χαίρομαι πολύ που είναι από τις προτεραιότητές σας. Έχουμε κείμενο εγκεκριμένο και είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε σε διαπραγματεύσει. Είμαι βεβαία λοιπόν ότι θα βρούμε πολλά σημεία που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί αυτό που επιθυμεί το Κοινοβούλιο και προέκυψε και από το κείμενο στην ψηφοφορία το πρωί είναι να δοθεί όθηση στην ε, ανάληψη αυτής της νέας μορφής μεταφορών, του συνδυασμού των τρόπων μεταφορών. Δηλαδή να περάσουν ε, τα μεγάλα φορτία και το μεγάλο βάρος από τους δρόμους και να πάει στους σιδηροδρόμους. Ε, πρέπει όμως να, υπάρχω, να υπάρχει και το ανάλογο ευρωπαϊκό δίκτυο για να γίνει αυτό. Ε, εγώ τώρα θα σας θυμίσω τον το τούνελ του Μπρένερο στις ε, ε, ένα θέμα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ιταλίας, γιατί πρέπει να παραμείνει ε, σε ροή η κυκλοφορία των εμπορευμάτων και το τούνελ του Πρένερο δεν ε, λειτουργεί αποτελεσματικά και θα πρέπει οπωσδήποτε να το φροντίσουμε για τα εμπορεύματα τουλάχιστον και να φροντίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει μετατόπιση στον σιδηρόδρομο και για το τούνελ αυτό και για την ε, σχέση με το πρώτο πακέτο κινητικότητας. Το καμποτάζ, την απόσπαση των εργαζομένων για το δικό μας το κείμενο όπως εγκρίθηκε, μπορούμε κάπως να ε, πούμε ότι βασιστήκαμε στα αποτελέσματα του πρώτου πακέτου τη κινητικότητας. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει, διότι χρειάζεται μια νομοθεσία αναφορά, μάλλον την νομοθεσία αναφορά την έχουμε ούτω ή άλλω. Ελπίζω λοιπόν από πλευρά Αυστριακής προεδρία να συνεργαστούμε αποτελεσματικά και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία Σμίτη για ένα λεπτό και επιστρέφω τον, ε, την Προεδρία στην ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ να σα καλωσορίσω θερμά κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ για τα όσα μα είπατε σήμερα εδώ. Αναφέρατε ότι ε, θεωρείτε πω η συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό βέβαια είναι πολύ ε, θετικό, αλλά υπάρχουν κάποια αδύναμα εντό εισαγωγικών ε, σημεία. Και αυτό για παράδειγμα συγκαταλέγεται το γεγονό ότι η Επιτροπή άφησε να παρέλθουν τρία χρόνια μέχρι τελικά να υποβάλει τι προτάσει τη για το πακέτο γενικότητα σε τρία τμήματα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και βέβαια τώρα ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να αντιμετωπίσουν 300 διαφορετικά ζητήματα πέραν του Brexit και πέραν ε, των υπολείπων ζητημάτων. Οπότε ε, πραγματικά έχουμε για πολύ, να κάνουμε πολύ μεγάλο αριθμό φακέλων και προτάσεων. Τώρα, Υπάρχουν μία σειρά από προτάσει, αλλά θα ήθελα ε, να αναφερθώ ειδικότερα στο ζήτημα των συνδυασμένων μεταφορών. Πραγματικά δηλαδή θα πρέπει εδώ τα όσα ε, ε, προτείνουμε να λάβουμε υπόψη μα ότι εξαρτώνται από τι χαμηλέ τιμέ, προκειμένου να υπάρχει και βιωσιμότητα αυτών των συνδυασμένων μεταφορών. Άρα λοιπόν τα όσα προτείνουμε εδώ μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο και το ερώτημά μου σχετικά είναι παρά του κοινωνικού πυλώνα, ο οποίο δεν πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα στο ε, στην Ολομέλεια θα κάνει περαιτέρω προσπάθειες ε, και μετά σε ό,τι αφορά την αυτοματοποιημένη οδήγηση ε, να πούμε ότι δεν έχει μόνο πλέον εκτήματα. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες περαιτέρω πτυχές σε ό,τι αφορά τους οδηγούς πίσω από την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Τι προβλέπετε να κάνετε ακριβώς. Ευχαριστούμε όλα. Προσπαθείτε να σέβεστε το χρόνο σας γιατί μετά άλλοι συνάδελφοι θα προλάβουν και δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Λουκασέφσκα. Κύριε Υπουργέ, θα είχατε την καλουσία να μας μιλήσετε για το συμβιβασμό, για το πακέτο κινητικότητας. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Ιδιαιτέρως προκειμένου να μην πληρώσουν την ύφη οι καταναλωτές, να μην κλείσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην φορτωθούν με γραφειοκρατία και έτσι ώστε οι μεταφορικές εταιρείε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα των ε, χωρών διαμετακόμισης. Στα, στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα πληρωμής διοδίων. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. και ποια θα είναι τα καθηγόντα της καινούριας ε, ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Απασχόλησης. Ευχαριστώ, Υπουργέ Χόφα. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Ε, σε ό,τι αφορά τη θέση σας, σε ό,τι αφορά την κατάργηση της αλλαγής του ωραρίου. Μετά, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των, της ε, μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, ε, τα ε, φορτηγά, τι ακριβώς θέλετε να κάνετε εδώ και σε ό,τι αφορά επίσης τους σιδηροδρόμους, ποιες είναι συγκεκριμένα οι προτάσεις σας. Είδατε ότι μόνο μισό λεπτό χρειάστηκε. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστούμε Υπουργέ. Κάθε Προεδρία φέρνει μαζί τη τα θέματα που ενδιαφέρουν πιο πολύ την κοινή γνώμη τη κάθε χώρα. Το είδαμε με την Εστονία και την ψηφιοποίηση, το είδαμε με τη Βουλγαρία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει, η Ευρώπη που προστατεύει, είναι ένα πρόγραμμα που φαίνεται να μα μιλάει για τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο οικονομικό, ε, ψηφιακό, για ανακύκλωση, για, ε, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, ναρκωτικά εμπορία ανθρώπων μας κάνετε να σκεφτούμε ότι στην Αυστρία τα πράγματα είναι τελείως εκτός ελέγχου. Όμως ε, για τα σύνορα της ε, Αυστρίας και για το Φριούλι, Βενέτσια, Τζούλια, την περιοχή, η περιφέρεια αυτή της Ιταλίας, ε, τι θα γίνει με τον Μπρένερο και τον Νταρβίζιο και Ποιε συνέπειε προβλέπετε για τι μεταφορέ και τον τουρισμό, και ω προ τον τουρισμό, πώ θα συμφιλειώσετε την πολιτική αυτή με, τον, με την πολιτική ξενοφοβία και κλεισίματο που έχετε καταγρα... διαγράψει. Ευχαριστούμε, κυρία Ντέμοντε. Κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, μίλησατε για τη στατική του Δούναβη. Πολύ σημαντικό θέμα. Η Αυστρία συντονίζει τον τομέα τους, ε, που σχολείται με, τις, ε, με το Δούναβι σε συνεργασία με άλλες χώρες. Όμως δεν υπάρχει πολύ ε, ε, πρόθεση από άλλες χώρες να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση τη εξασφάλισης του ότι ο Δούναμις θα είναι πλωτός. Θα μπορέσετε να κάνετε κάτι έτσι ώστε οι χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Δούναμις θα χρηματοδοτήσουν το πλωτό του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντερσον, έχει το λόγο. Η Καρολίνα Γκράς δυστυχώς χρειάζεται να πάει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αλλά ζητά συγγνώμη. Δύο θέματα ήθελα να θίξει. Είπατε κάποια καλά λόγια για την προστασία των πολιτών και των αναζωμένων. Όμως, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης, θα μπορούσατε να μας πείτε τι θα κάνετε για να προχωρήσει το θέμα. Δεύτερον, να συμφωνήσω με τον κύριο Κράμερ για τη σημασία της ίσης πληρωμής των τομέα των μεταφορών και γενικότερα οι συνθήκες που επικρατούν στους παρόχους υπηρεσία θα, ε, θα πρέπει να ε, διορθωθούν. Ε, Επίση, θα πρέπει να δούμε το θέμα των δικαιωμάτων επιβατών, επιβατών στους σιδηροδρόμους, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και τη εφαρμογή εφαρμογής τους. Ευχαριστώ κ. Ζωτόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας ε, καλωσορίσω εδώ για την ανάληψη αυτού του καθήκοντος, του νέου καθήκοντος για σας ως πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα στα πολωνικά. dumping Dumping, Το κοινωνικό dumping είναι μια πρακτική που συνεπάγεται μια πώληση σε τιμή μικρότερη του κόστους. Ε, μια ε, πώληση αγαθών αλλά και υπηρεσιών. Το dumping είναι αρνητικό Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ακριβώς ορίζετε ως κοινωνικό ντάμπινγκ εσείς. Και μετά αν μιλάμε για ίδια πληρωμή, για ίδια εργασία, γιατί δεν λέμε ίδια εργασία, ε, ίδια αμοιβή στον ίδιο εργοδότη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αρνοτού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε Υπουργέ που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε και για την ομιλία σας. Είπατε ότι η προτεραιότητά σας θα είναι να προστατεύετε καλύτερα, γιατί τέτοια προτεραιότητα έχουμε και εμείς. Και συμφωνώ απολύτως. Να προστατεύσουμε τους πολίτες των κρατών μελών, να προστατεύσουμε τους συμπολίτε μας, αλλά και τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας. Σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης, εντατική που καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και ο τομέα τη αεροπλοεία είναι επίση σημαντικό. Μια ε, συνεδρία σε υψηλό επίπεδο θα γίνει στη Βιέννη τον Οκτώβριο για το θέμα αυτό, ε, υπό την αιγίδα τη Προεδρία σα. Και ακόμα υπάρχουν σοβαρέ αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών. Οι αεροπορικέ εταιρείε και οι διάφοροι φορεί στην αεροπλοεία, ανάλογα με το αν ε, ασχολούνται με τα αεροσκάφη και την Airbus, με τι ε, χερσαίε επιχειρήσει ε, ή με οποιοδήποτε άλλο κλάδο τη βιομηχανία, έχουν και διαφορετική θέση. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε τι σκοπεύει να προωθήσει η Αυστρία ω θέση σε αυτή την σύνοδο και τι περιμένετε να προκύψει ω αποτέλεσμα. Τι θα γίνει για να έχουμε ισότιμε ε, προποθέσει για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, των οποίων η θέση απειλείται από τι εταιρείε του κόλπου, των κρατών του κόλπου, του αραβικού κόλπου κυρίω. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, σωρία ερωτήσεων, σωρία και απαντήσεων. Θα σας δώσουμε το χρόνο για να απαντήσετε σε όλες και αν χρειαστούν διευκρινήσεις θα φροντίσουμε να τις ζητήσουμε από τους συνεργάτες σας. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στο σύνολο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Και μην ξεχάσετε να μας, και μην ξεχάσετε να μας πείτε και τι μέθοδος είναι αυτή του κογκλαβίου, αυτών των συνδυασμών που θα χρησιμοποιήσετε. Ναι, να σας ε, πω ότι σε ό,τι αφορά τα πακέτα κινητικότητας, τουλάχιστον σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο ε, πακέτο, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ απόψεων και για παράδειγμα εντό ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και άρα λοιπόν σκέφτηκα Πώ θα μπορούσαμε να γεφυρώσουμε τα χάσματα ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Σκέφτηκα λοιπόν να έχουμε εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν τις, τη μεγαλύτερη διάσταση απόψεων μεταξύ τους ε, προκειμένου ε, ε, να, να, να, να, έρθουν λοιπόν σε αυτά τα κονκλάβ, σε αυτές τις συναντήσεις εκπρόσωποι από αυτές τις χώρες με ιδιαίτερες διαφορές απόψεων προκειμένου να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή αυτών των απόψεών του ε, και προκειμένου δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια προτού πούμε απλώ και μόνο ότι αποτύχαμε ευθύ εξ αρχή. Τώρα, αξιότιμε ε, κύριε Βαντεκάμπ, θα ήθελα καταρχήν να σα ευχαριστήσω για, τις, ε, για τα συγχαρητήριά σα για την ανάλυση τη Προεδρία. Ε, μας είπατε ότι ε, οι πιο ηλικιωμένοι δεν θα έπρεπε να έχουν επικίνδυνα σπορ, έτσι, και επειδή εγώ ήμουν ε, μεστέχνης ε, πιλότος, εντάξει, εμ, μπορώ να σας πω ότι πράγματι με τα χρόνια έχω γίνει πιο προσεκτικός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πράγματι έχουμε να κάνουμε εδώ με δύο πολύ ισχυρούς παίκτες εντό εισαγωγικών και βέβαια δεν γνωρίζω πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα στις ΗΠΑ με τον προστατευτισμό. Σε ό,τι αφορά την Κίνα γνωρίζουμε πώ ε, θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα είναι δηλαδή ο πιο σημαντικό οικονομικό πόλο ε, του κόσμου στο μέλλον, με τη μεγαλύτερη τουλάχιστον αγοραστική δύναμη, οπότε θα πρέπει να βρισκόμαστε και να διατηρήσουμε καλέ φιλικέ ε, σχέσει απέναντι στην Κίνα, απέναντι στι ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντά μα. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σε ό,τι αφορά του σημαντικού τομεί να συνεργαζόμαστε μεταξύ μα. Τώρα, αναφερθήκατε στο ζήτημα των διοδίων. Και τέθηκε επανειλημμένα αυτό το ερώτημα. Ε, και εδώ αναφέρομαι δηλαδή στα διόδια σε ό,τι αφορά επιβατικά έως 3,5 τόν. Εδώ έχουμε τα διαφορετικά κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τα διαφορετικά τους εθνικά συστήματα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ε, ένα φόρο πετρελαίου, δηλαδή ε, έχουμε τον κανονικό φόρο ε, στον οποίο προστίθεται για παράδειγμα ένα τέλος σε ό,τι αφορά κάθε λίτρο πετρελαίου ή βενζίνης και αυτό βέβαια με, την, ε, με τη σειρά του έχει μια επίπτωση ε, στον τρόπο οδήγησης γιατί αν οδηγώ πιο ήπια τότε φυσικά η κατανάλωση είναι λιγότερη και κατά συνέπεια και το σχετικό τέλος. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς είναι διαμορφωμένα τα διαφορετικά εθνικά συστήματα επιβολής τελών διοδίων. Πάντω, όπω σα είπα, σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε έστω και μέσα τη δική μα ε, θέση. Ε, τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το, τον προπολογισμό, βέβαια πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά κυρίω το, το ε, Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ο καγκελάριό μα πράγματι σωστά το είπατε, πω θέλει εδώ να έχει να κάνει κάποιε οικονομίε. Αλλά ποιοι είναι οι βασικοί τομεί στου οποίου θα πρέπει να εστιάσουμε. Οι συνδέσει ε, στι μεταφορέ ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέσει ευρυζωνικέ, διαδικτυακέ, εκπαίδευση. Αυτοί λοιπόν είναι οι τιμέ στου οποίου έχουμε ιδιαίτερη, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα και σε σχέση με αυτού του τομεί θα πρέπει ο προπολογισμό να είναι κατάλληλα πληκοδοτημένο. Τώρα, αναφερθήκατε στο ζήτημα των λιμένων εσωτερική ναυσιπλοεία και πράγματι ε, εδώ το, το, έχει πολύ σημαντικό ρόλο και το, το project των ε, χωρών του δρόμου του μεταξιού γιατί εδώ θα δημιουργηθούν κάποια hub, κάποιοι, κάποια κέντρα αν θέλετε διέλευσης τα οποία καλό θα είναι να δημιουργηθούν ε, και σε λιμένες και σε αερολιμένες έτσι ώστε να μην δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και πάλι στο πλαίσιο αυτού του δρόμου να μην δοθεί δηλαδή όλη η έμφαση στις οδικές μεταφορές. Ε, ζητώ συγγνώμη για τη βραχνή φωνή μου. Ακούγομαι λίγο σαν τον Τζο και το γνωρίζω, αλλά ε, κάτι κόλλησα κάπου. Τώρα. Ε, μου θέσατε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους στόχους της Αυστριακής Προεδρίας. Σας ε, λέω ότι πραγματικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε πρόοδο σε σχέση με τα διαφορετικά και οι συνεργάτες μας ήδη έχουν ξεκινήσει ε, μία σειρά από επαφές, επαφές προκειμένου να φτάσουμε Έχουμε ξεκινήσει επαφές για να φτάσουμε σε συμβασμού και θα υπάρξουν 150 συνολικά συνεδριάσει ομάδων εργασία του Συμβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα υπό την Προεδρία μα. Τώρα, αναφέρθηκε και το ζήτημα των δίκαιων κοινωνικών συνθήκων. Έχουμε το Road Alliance ε, και άλλα, για παράδειγμα. Αυτό το ζήτημα τη ε, καμπίνας ε, του οδηγού. σε σχέση με αυτό νομίζω πω μπορούμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό εάν καταφέρουμε ε, πράγματι το να διασφαλίσουμε ότι οι οδηγοί φτάνουν στην ώρα του στο σπίτι του. Γιατί πολλοί οδηγοί μα λένε ότι τελικά καταλήγουν στο να κοιμούνται σε ένα ξενοδοχείο ή οπουδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να επιτύχουμε εδώ ένα αποτέλεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό dumping, ε, αναφέρθηκε και το ζήτημα των 12 ωρών εργασία ε, ανά ημέρα. Εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα για την πλευρά τη Προεδρία. Ε, είναι αυτονόητο έχει αποφασιστεί ότι δηλαδή ανά ημέρα θα πρέπει το μέγιστο όριο ωρών εργασία να είναι οι 12 βασιζόμενοι πάντοτε στην κανονική, στο κανονικό οργάνιο εργασίας των 8 ώρων και 40 ημερών ανά εβδομάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, τον Μπρένα τώρα που αναφέρθηκε εδώ, ναι, πράγματι βρισκόμαστε σε προπαρασκευή ε, του σχετικού άξονα, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες ε, ε αρτηρίες που οδηγούν εκεί. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου συγκεκριμένη διέλευση να αποσυμφορηθεί και θα πρέπει βέβαια ε, οι λύσει που θα εφαρμόσουμε εδώ να είναι ε, δίκαιε. Πάντω, σε ό,τι αφορά αυτό το τρίγωνο των τούνελ, αν θέλετε, προφανώ δεν είναι τόσο εύκολο να. Ε, επιτύχουμε πρόοδο από τη μία μέρα στην άλλη. Πάντως ε, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή ε, που εστιάζουμε είναι οι οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκεί στον Πρένα. Τώρα, αναφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας από διάφορους βουλευτές. Προφανώς θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό ζήτημα για αυτή την αρχή και οι κοινωνικές συνθήκες στον τομέα των μεταφορών. Και εδώ μπορεί, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που ενεργούνται στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε και να αναμείνουμε το τι θα κάνει η αρχή αυτή σε αυτό το τομέα. Μπορούμε ήδη να αναλάβουμε δράση από την δική μας πλευρά. Νομίζω ο Βουλευτής Τσίλε έθεσε ένα ερώτημα για να τον τοποκάστε. Συγγνώμη. Ε, αναφέρθηκε λοιπόν ο βουλευτής ε, Τσίλε στο σύνθημά μας, στο μια Ευρώπη η οποία προστατεύει και ότι σε σχέση με αυτό το ζήτημα της ασφάλειας της μεταφοράς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ό,τι αφορά λοιπόν τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Ε, ορισμένα μέλη λοιπόν του Συμβουλίου θεωρούν ε, είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό το ζήτημα σε συνάρτηση με το ζήτημα της πρόσβασης στην εργασία και της πρόσβασης ε, στην αγορά ε, μεταφορών. Ε, σε σχέση λοιπόν με αυτό το ζήτημα συνεχίζεται η συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα και θα πρέπει ωστόσο να σας πω ότι προτεραιότητα δίνουμε στο να επιτευχθεί πρόοδο σε ό,τι αφορά τι κοινωνικέ συνθήκε στο πλαίσιο του πακέτου κινητικότητα. Αναφέρθηκε επίση για το ζήτημα των διασυνοριακών μεταφορών. Εδώ έχουμε ξεκινήσει ήδη κάποιε διαβουλεύσει και ε, πράγματι βλέπουμε ότι εδώ μπορεί να υπάρξει αντίκτυπος και στο επίπεδο της περιφερειακής και τοπικής ε, πολιτικής ε, ε, κινητικότητας και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει εντατικές διαπραγματεύσεις. Πολλά κράτη-μέλη θεωρούν πως υπάρχει εδώ όμως μία απειλή για την, αρχή της, την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Άρα λοιπόν το να κλείσουμε τι διαβουλεύσει στο πλαίσιο τη Αυστριακή Προεδρία για αυτό το πακέτο κινητικότητα το θεωρώ κάπω δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των ενόπλων δυνάμεων, ε, το Ομοσπονδιακό ε, Υπουργείο για την Ευρώπη, την ολοκλήρωση και ε, τα σχετικά ζητήματα είναι το αρμόδιο. Πάντως, σε στενή συνεννόηση με άλλους ε, συναρμόδιους ε, φορείς ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα και από, από ειδικότερα από την πλευρά του δικού μας Υπουργείου εστιάζουμε στο ζήτημα της συμβατότητας της σχετικής υποδομής για την κινητικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου ε, θα πρέπει όλες αυτές οι εργασίες εδώ να συνεχιστούν λαμβάνω, σεβόμενοι πλήρως τις σχετικές ε, τις αρμοδιότητες και την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών ε, σεβόμενοι επίσης και την τεχνική ουδετερότητα και ε, ε ευθυγραμμίζοντας αν θέλετε τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων μεταφορά στρατιωτικής και μη στρατιωτικής χρήσης. Τώρα ο κύριος Τέλετσκα με ρώτησε ή μάλλον τοποθετήθηκε σχετικά ότι ε, η Αυστρία έχει παραδοσιακά μια πολύ καλή αίσθηση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ειλικρινή διαμεσολαβητή. Ε, πραγματικά να το επαναλάβω αυτό και να σας το υποσχεθώ ότι θα το κάνουμε. Ε, πραγματικά ο ανταγωνισμός στον οποίο βρισκόμαστε εκτεθειμένοι ως Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για μας όλους μας να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Και σε αυτό το πλαίσιο τίθεται το και το, το σχετικό ζήτημα του ότι δηλαδή βλέπουμε τις υπομετρήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο είναι οικονοποιημένοι οι πολίτες μας Βλέπουμε λοιπόν το ότι να τίθεται το ζήτημα του τι είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα απόμακρο φορέα κάπου μακριά, είναι και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και δεν θα πρέπει δηλαδή κανεί απλώ να ε, μεταβάζει ουσιαστικά, να μετακυλεί την ευθύνη για όλα τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν υπάρχουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι αυτό οφείλεται στι αποφάσει που λαμβάνουν οι πολιτικοί των επιμέρου κρατών μελών. Δεν είναι αποφάσει που λαμβάνει ένα απόμακρο ε, φορέα στι Βρυξέλλε. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μα έχουμε την ευθύνη ε, για να συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά ζητήματα. Και νομίζω πω εδώ πρόκειται για ε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, έχει επικουρικό ακριβώς χαρακτήρα, όπου δηλαδή τα βασικά προβλήματα εθνικού χαρακτήρα λύνονται από τα εθνικά κράτη, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν ζητήματα διεθνή, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν με μόνο μένα τα κράτη-μέλη. Μετά. Όταν τώρα κανείς μπερδεύει τα χαρτιά του, όπως το έκανα εγώ μόλις τώρα, τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Κάντε λίγη υπομονή. Abgeordneter Kramer, warten Sie, ich schau mal. Sie sind nicht böse, wenn ich mit der Frau Abgeordneten Ναι. Ε, κύριε Κράμερ, ε, θα σα θα σας απαντήσω και εσά. Εν πάση περιπτώσει, καταρχήν να απαντήσω στο ζήτημα των ε, συνδυασμένων μεταφορών. Και το Μπρένα και πάλι. νομίζω πω ο Μπρένα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου οι μεταφορές να περάσουν στο σιδηρόδρομο. Ε, γνωρίζουμε και αυτήν την ε, φέβρεση, την νεκράζα, ε, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την μετάβαση από το, τις οδικές συνδρομικές μεταφορές και ακριβώς σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στην αποσυμφόρηση του Τενεραμπρένα ώστε να έχουμε περισσότερο σιδηρόδρομο εκεί. Ε, έως το 2027 θα έχουμε ολοκληρώσει το σχετικό ε, αυτό το έργο και βέβαια έχουμε επενδύσει 13,9 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό το σε αυτό το έργο το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ ψηλό ποσό για ένα μικρό κρατός μέρος όπως ε, εμείς. Ε. Τώρα, ο... η ε, Ευρωβουλευτή Σμίτα αναφέρθηκε στο ζήτημα το ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία που έχουμε διοργανικά και αναφερθήκατε και στις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις που έχουμε στο πλαίσιο του Brexit. Οι εξελίξεις βέβαια και η κατάσταση για την Προεδρία μας έγινε πιο δύσκολη μέσω ακριβώς ε, του Brexit, ειδικότερα σε ό,τι αφορά και το μέλλον ε, των ε, μεταφορών και το τι θα ακολουθήσει. Γιατί αυτό που θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου είναι ότι ναι, μεν αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν αποχωρεί από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό μα εταίρο σε ό,τι αφορά ζητήματα ψηφιοποίηση, περαιτέρω εξέλιξη των μεταφορών και ούτω καθεξή. Άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθο να πούμε στο Ηνωμένο το εξή αποχωρήσατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα θα κάνουμε τη ζωή σας όσο πιο δύσκολη γίνεται. Όχι, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ε, και επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, πραγματικά τα, αυτή τη στιγμή ήδη μεταβιβάζουμε τεράστιο όγκο δεδομένο και για τα αυτόματα οχήματα θα είναι ακόμα ε, πιο αυτοματοποιημένα. Και θα δούμε τι, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα δεδομένα και έχει γίνει και μια σχετική διαβούλευση ε, στη Βιέννη για αυτό το ζήτημα. Τώρα, ε, κυρία Περεύσκα, αναφέρθηκε στο ζήτημα του κόστου που θα προκύψει για του καταναλωτέ από το πακέτο κινητικότητα. Προφανώ το ζητούμενο εδώ να διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο τι διατάξει που να μην οδηγήσουν σε ε, περισσότερη επιβάρυνση, σε περισσότερη γραφειοκρατία. Ε, πρόκειται για ένα κοινό μα στόχο και αν καταφέρουμε να επιτύχουμε ε, ε, μία προσέγγιση ανάμεσα στα Borderlands και στα, στις, στα, στις χώρες του Βίζεγκρατ. Καλό είναι ε, να, το, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί. Γιατί ε, τα κράτη-μέλη από μόνο τους περιπλέκουν τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιπλέκει και αυτή από δική τη πλευρά τα πράγματα, οπότε σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο πακέτο θα πρέπει ε, να μην περιπλακούν περισσότερο τα πράγματα, γιατί τελικά πάντοτε σε όλες τις προτάσει εκείνος που ε, καταβάλει το κόστος του είναι ο τελικό καταναλωτής. Τώρα, ο ε, βουλευτής Κοχ έθεσε ένα ερώτημα σε σχέση ε, με το Ecoliner και και το ότι αποτελεί μια πολύ ωραία έννοια ή το Monster Trucks ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ανάλογα με το ποιος, ε, ε, τι πρόσβαση έχει κανείς. Ε, δηλαδή έχω ένα όχημα το οποίο αν το χρησιμοποιώ έχω χαμηλότερες εκπαμπές κατά 35% ωστόσο με την, με την αλλαγή στο σιδηρόδρομο ουσιαστικά ε, είναι η προτιμητέα επιλογή γιατί αν ε, επιλέξω και πάλι ε, οδική μεταφορά ως εναλλακτική ουσιαστικά πάλι αυξάνω τον ανταγωνισμό στον οποίο βρίσκεται εκτεθειμένος ο σιδηρόδρομος. Οπότε αντιλαμβάνομαι την απέτηση εδώ, την αξίωση από την πλευρά του, του, κλάδου των μεταφορών αλλά η, η δική μου προσέγγιση είναι Α μεταβιβάσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι των περιβαλλοντικών μεταφορών στο σιδηρόδρομο. Γιατί έχουμε επενδύσει και στο επίπεδο τη κινητικότητας εκεί, οπότε θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε τα πράγματα και νομίζω πω ε, αυτό το Giga το Ecoliner και το τα γενικά η σχετική πρόταση έχει απορριφθεί και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δούμε λοιπόν ε, πώ μπορούμε εδώ να αυξήσουμε για παράδειγμα και την ενδεχομένω την κινητικότητα με βάση το υδρογόνο και το καθεξή. Ε, τώρα, η, ε, αναφέρθηκε το ζήτημα και πάλι της ε, θερινής περίοδου και το ότι ε, έχει υποβληθεί με πρόταση από την πλευρά ε, προς, προς την Επιτροπή και σε ό,τι αφορά δηλαδή το, το, το θερινό ωράριο και την αλλαγή που γίνεται εδώ είχε υποβληθεί μια σχετική πρόταση και εγώ είμαι προσωπικά υπέρ. Τώρα, ο, ε, κύριος Κράμερ αναφέρθηκε στο ζήτημα της επιβολής της ε, γερμανικής, ε, των γερμανικών διοδίων και της προσφυγής που έχει γίνει. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορεί να αρθεί αυτή η προσφυγή, αλλά αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση που θα εκδώσει το δικαστήριο. Ε, αντιλαμβάνομαι γιατί επιβάλλει αυτά τα διόδια η Γερμανία. Πάντως, Δηλαδή επιβάλλει μια επιβάρυνση αλλά απαλλάσσει από αυτή την επιβάρυνση τους ε, Γερμανούς πολίτες. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε πολλούς άλλους τομείς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οδηγούσε τελικά σε μείωση της αλληλεγγύης, σε ένα κατακαιρματισμό αν θέλετε. Ε, οπότε της, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική στη, λογική, αν θέλετε, αυτή τη πρόταση τη Γερμανία. Αντιλαμβάνομαι τη λογική σε ό,τι αφορά τα διόδια, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει μια τέτοια αρχή, ότι δηλαδή επιβάλλω ένα τέλο, το οποίο όμω δεν ισχύει για του δικού μου πολίτε. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν είναι, είναι προβληματική. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αναφέρθηκε από τον ε, κύριο Κράμερ εκτό μικροφώνου. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν το τομέα των ε, σιδηροδρόμων, για... από, από το Ζόμπατα για παράδειγμα, μέσω Όμπερβαρτ, με τελικό προορισμό το Ρίχτμπεργκ. Είχαμε για παράδειγμα, σας αναφέρω αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική στο, στο παρελθόν, αλλά με τις ε, δύο παγκόσμιους ε, πολέμους ουσιαστικά δεν καταργήθηκε αυτή η ε, σύνδεση και τώρα γίνονται συζητήσεις προκειμένου να επανενεργοποιηθεί αυτή η σιδηροδρομική γραμμή γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική αρτηρία για μεταφορές και βέβαια ήδη σας είπα ότι προσπαθούμε να επενδύσουμε πολλά κονδύλια σε αυτό το τομέα της σιδηροδρόμων δηλαδή μεγάλων αποστάσεων τώρα. Αναφέρθηκε ότι λόγω του σλόγγαν που επιτύχαμε, ε, που, που επιλέξαμε μάλλον ως Αυστριακή ε, Προεδρία, ότι η κατάσταση στη χώρα μας είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Ε, αυτό το σύνθημα δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε ένα, μια Ευρώπη η οποία περιχαρακώνεται. Όχι, αυτό που εννοούμε με αυτό το σύνθημα είναι ότι όταν θέλουμε να προστατεύσουμε το χώρο Σέγγεν, να εξετάσουμε ποιο διέρχεται τα σύνορα του χώρου Σέγγεν. Αυτό λέμε προστατεύουμε ε, τα σύνορα. Αλλά και βέβαια το, η Ευρώπη που προστατεύει σημαίνει και ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών. Δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η αρχή σε όλου του τομεί. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιχαρακωθεί. Όχι, θα πρέπει να διασυνδεθεί περισσότερο. Και για παράδειγμα στο επίπεδο τη ψηφιοποίηση. Αναφερόμαστε και στο ζήτημα για παράδειγμα τη διαστημική έρευνα. Άρα λοιπόν θέλουμε μια ανοιχτή Ευρώπη η οποία όμω γνωρίζει τι πιέσει τι οποίε βρίσκεται εκτεθειμένη έξω. Γνωρίζετε για παράδειγμα ότι υπάρχουν τρομοκράτε οι οποίοι έχουν προβεί σε παχθέστατε ε, πράξει οι οποίοι έχουν καταφέρει ακριβώς αξιοποιώντας ε, την, ε, το άσυλο να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς γιατί ε, ισχυρίστηκαν ότι χρειάζονταν προστασία. Οπότε ακριβώ θα πρέπει να δούμε ποιο πραγματικά χρειάζεται προστασία και άσυλο. Τώρα, αναφέρθηκε ή ζητήθηκε ε, να πούμε ποια είναι η στρατηγική των ε, κρατών μελών από τα οποία ε, διέρχεται ο Δούναβης. Είπαμε ότι θα υπάρξει και αυτή η συνάντηση των σχετικών κρατών και εδώ η σχετική ναυσιπλοεία στο Δούναβη που μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μια σημαντική συμβολή στις πολιτικές μεταφορές, αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα διασφαλίσουμε το ότι, είναι, ε, ότι μπορεί να, ε, είναι δυνατή η ναυσιπλοεία σε όλα τα τμήματα του Δούναβη. Γιατί αν υπάρχει σε, ένα, σε μια χώρα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ναυσιπλοεία στο Δούναβη, ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρχει ναυσιπλοεία στο σύνολό του. Υπουργέ, θα σα παρακαλέσουμε να ολοκληρώσετε, γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα δυστυχώ μιλήσει για διαταξή μα. Υπάρχει επόμενο θέμα. Εάν μπορείτε σε ένα λεπτάκι κάπως να τα ε, πείτε όλα, γιατί έχουμε και άλλα σημεία και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να ξανασυζητήσουμε σε κάτι που ανέφερθηκε από σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ε, των μεταφορών και τις συνδυασμένες μεταφορές. Ε, πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για την Αυστριακή Προεδρία. Ζητώ συγγνώμη που δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Μπορούμε να υποβάλουμε γραπτώ κάποιε απαντήσει. Ε, ήταν ενδιαφέροντα τα ερωτήματα. Πάντω, να πω ε, κλείνοντα ε, πω για μα η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι επιτροπέ είναι πολύ σημαντική για μα. Εγώ ήμουν εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου εδώ στην Αυστρία για 6 μήνε, οπότε γνωρίζω πω μπορούμε να φτάσουμε σε κοινέ λύσει και θα ήθελα πραγματικά να σα προσκαλέσω να κάνετε το εξή. Εάν έχετε την αίσθηση ότι ακολουθούμε μία λανθασμένη κατεύθυνση από την πλευρά τη Προεδρία μα σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα, να έρθετε άμεσα σε επαφή μαζί μου ε, προσωπικά. Γιατί πραγματικά θέλω να βρούμε κοινέ λύσει για την Ευρώπη μα και για αυτή την κοινή μα ε, πατρίδα, αν θέλετε, την Ευρώπη. Και σα ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Αν όταν δεν είμαστε σύμφωνοι μαζί σας, το που λέμε, γιατί και εσείς είστε πολύ ειλικρινείς μαζί μας. Μίλησατε για τις προτεραιότητές σας, ε, για την κινητικότητα. Υπάρχουν κλιματολογικά, ενεργειακά θέματα, θέματα οδικής ασφάλειας. Οπότε τώρα ας σηκώσουμε τα μανίκια και ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε θα θυμάμαι πάντα αυτό που λέτε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στον κόσμο και θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη Ευρώπη για μια Ευρώπη που προστατεύει. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ξαναρχίζουμε. Κύριε Ρότερς, Ελάτε, παρακαλώ πολύ, ελάτε μαζί μου. Μη, φο... μη με φοβάστε. Alors, le prochain point à l'ordre du jour. Επόμενο σημείο της μέσης διάταξης παρουσίαση από την Κομισιόν της πρότασης για τον μηχανισμό διασύνδεσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Στόχος είναι η Επιτροπή μας να ενημερωθεί για το μέλλον της Επιτροπής, του, του Μηχανισμού Διασύνδεσης και πώς αυτός εντάσσεται στην, ε, στην πολιτική διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. η συζήτηση θα συνεχίσει ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή με την οποία μάλιστα θα συναντηθούμε από κοινού για να επεξεργαστούμε μια κοινή θέση για την προετοιμασία του μηχανισμού διασύνδεσης για όλη την ε, για τις μεταφορές αλλά και για την ενέργεια και το ψηφιακό μαζί. Καλώς ήρθατε ξανά, λυπάμαι πολύ που έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ε, έχετε έξι λεπτά λοιπόν. έτσι ώστε οι εισηγητέ μα να προλάβουν να λάβουν το λόγο. Και ο Στέλσκα και ο κ. Μαρινέσκου θα επανέλθουν σύντομα, είμαι σίγουρο. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας για την, επιτροπή μας, ε, για την, για την πρότασή μας που είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε πράγματι μπορώ να είμαι πιο σύντομο, θα εστιάσω στα πιο βασικά και θα μιλήσω στα αγγλικά, αν, μου επιτρέπετε. Ορισμένα σημεία κλειδιά λοιπόν. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε την πρόταση της ε, Κομισιόν για την ε, διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, που είναι η συνέχεια της ε, υφιστάμενης γνωρίζουμε πολύ καλά την, τον κανονισμό του, των διευρωπαϊκών δικτύων και για την, και τις διευκόλυνσης στην Ευρώπη. Αυτή πρόκειται για τη δεύτερη τέτοιου είδους πρωτοβουλία ε, και για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Στα πάνω αριστερά βλέπετε τις τρεις ε, ε, γραμμές του προπολογισμού που αφορούν ε, την, διαδικα... την αυτή. Έχουμε όμως και άλλους προπολογισμούς που έχουν για την εφαρμογή του, ε, των ευρωπαϊκών δικτύων, όπως βλέπετε. Επόμενη διαφάνεια. ορισμένα σημαντικά θέματα Τα βασικά θέματα ξέρετε ήδη βέβαια. Είχαμε κάποια εισαγωγικά, τα πέρασα για να εστιάσουμε στα επόμενα. Καταρχήν προτείναμε να ε, κατανείμουμε στα 60-40 τον προπολισμό, το 60% για το, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το 40% για, τον, ε, για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου και το δεύτερο ε, για τη λειτουργία. Το 60% ε, ε, ε, αφιερώνεται στο, κατά 75% στο κεντρικό δίκτυο και το υπόλοιπο για, για τους διαδρόμους μάλλον το 10% για τα υπόλοιπα κομμάτια του κεντρικού δικτύου και το 15% για το υπόλοιπο κομμάτι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί φτάνει το 2000, στο 2015 το 2050 και θα πρέπει να εφαρμόσουμε, να υλοποιήσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια, όχι μόνο το κεντρικό δίκτυο. Το 40% είναι πολύ σημαντικό όμως, που αφορά τον εξυγχρονισμό ε, του, του, του υπάρχοντος δικτύου και αφορά ε, όλες τις εφαρμογές για παράδειγμα το Cesar και το VTMIS, το ERTMS, συγγνώμη. Το ERTMS δεν περιορίζεται στο κεντρικό δίκτυο. Αφορά το σύνολο του δικτύου. Εδώ θα έχουμε και προγράμματα διαλειτουργικότητας, ασφάλεια, οδικής ασφάλειας κλπ. Δεν μπορούμε αυτά να τα περιορίσουμε στο κεντρικό δίκτυο. 60% και 40% λοιπόν σε αυτούς τους δύο πυλώνες. Ε, σκοπίμως για να καλύψουμε και τις βασικές υποδομές ως πρώτη προτεραιότητα, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συνολικού δικτύου. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε την στερεωτική κινητικότητα. Θα με ρωτήσετε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό. Στο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνεται η στερεωτική κινητικότητα ε, Κατά τη διάρκεια των επόμενων Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα καθοριστούν οι στρατιωτικές απαιτήσει. Έτσι ώστε θα εντοπίσουμε τις διαφορές, τα κενά που έχουμε ανάμεσα στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα. Και θα εντοπίσουμε τις, υποδομές, τις διτές υποδομές που χρειάζονται. Δεν θέλουμε να έχουμε μόνο αποκλειστικά ε, στρατιωτικές υποδομές. Οπότε οποιοδήποτε επενδύσεις σε αυτό το, από αυτόν τον προπολογισμό περιορίζεται στο στα ευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορών. Δεύτερον, αυτό ο προπολογισμό θα υλοποιηθεί μέσω της διευκόλυνση σύνδεδος στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε δύο πράγματα. Περιορισμός στο, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Δεύτερον, χρησιμοποίηση της ε, δια, ε, στην Ευρώπη. Μέσω project διπλή χρήση. διότι ε, δεν θα λοιπόν πολύ, δεν θα ακούσουμε πολύ στο μέλλον τη χρήση από στρατιωτικές μονάδες αυτών των υποδομών, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αναπτύξουμε τέτοιου είδους υποδομές. Δεύτερη, ε, επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε πάλι τους τρεις προϋπολογισμούς της ε, διευκόλυνσης στην Ευρώπη. Γενικό προϋπολογισμό, ε, στρατιωτική κινητικότητα και ε, συνοχή. Και έχουμε και, και μια σύγκριση με τη σημερινή περίοδο. Η, στη νέα αυτή διευκόλυνση προτείνουμε να μην ε, το 100% σε εθνικούς φακέλους, αλλά το 70% και το υπόλοιπο 30% να είναι διαθέσιμο με ανταγωνιστικά κριτήρια αν όλα τα δίναμε σε, με βάση ανταγωνιστικά κριτήρια, τότε θα είχαμε μόνο διασυνοριακά project, ενώ εμείς θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο και τα θέματα συνοχής. Νομίζουμε ότι όλες οι χώρες συνοχής έχουν τέτοια project, για παράδειγμα Δούναβη, ε, σιδηροδρομικές συνδέσεις, λιμενικές συνδέσεις κλπ. Και θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο προβλέπουμε ότι όχι μόνο μετά τα πρώτα τρία χρόνια θα δίνουμε project, ε, χρηματοδότηση με ανταγωνιστικά κριτήρια, αλλά από την αρχή. Έτσι θα ενισχύσουμε την, το όραμα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και τη συνοχή στο μέλλον της Ευρώπης. Τελευταία μου διαφάνεια. Ε, συντελεστές συγχρηματοδότησης, ποσοστά συγχρηματοδότησης. Και εδώ έχουμε μια αλλαγή, πηγαίνουμε στο 50% τα διασυνοριακά στο γενικό προπολογισμό και 85% σε ό,τι τα κονδύλια της συνοχής. Αυτό είναι σημαντικό διότι τα ποσά της συνοχής είχαν ως τώρα 70% συγχρηματοδότηση και πολλά από αυτά τα project θα ολοκληρωθούν με αυτό το ποσοστό. Για το γενικό προϋπολογισμό, το 30 το πήγαμε στο 50. Ε, δεν θα μιλήσω για την γεωγραφική κατανομή. Ε, τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο, να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μαρινέσκου. Ο λόγος εσάς για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Νομίζω κάποιες από τις θέσεις μου τις ξέρετε. Απλώς ένα γενικό σχόλιο Μπορείτε να κάνετε τα πάντα τώρα. Μπορείτε να πάτε τη χρηματοδότηση εκεί που θέλετε. Μέσω των προγραμμάτων μας. Μέσω της υλοποίηση. Το κοινοβούλιο δεν έχει τίποτα να πει. Και εσείς θα επιλέγετε και τα έργα. Διότι μέσω του προγράμματος εργασιών θα λέτε τι είδους προγράμματα, τι είδους έργα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε. Αυτό το σχόλιο είναι γενικότερο. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Διότι μιλάμε για ε, ελεύθερο ανταγωνισμό. Για ποιον ελεύθερο ανταγωνισμό όταν εσείς αποφασίζετε πού θα πάει το χρήμα. Διότι η πραγματικότητα για όλα τα ποσά είναι η ίδια. Μετά για την κινητικότητα. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι η θεατρική κινητικότητα, η κινητικότητα των ενόπλων δυνάμεων είναι 6,5 δις. Και τα υπόλοιπα είναι 23 Νομίζω ότι ένα τέταρτο 20% ενός προγράμματος πρέπει να πηγαίνει για στρατιωτικούς σκοπούς. Να το σκεφτούμε και αυτό, γιατί στην εν λόγω περίπτωση πολλά προγράμματα θα έχουν να κάνουν με τα στρατιωτικά αλλά ένα 30 70% θα πρέπει από τη συνοχή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορείτε να... Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φτώχεια κάποιων κρατών ε, παίρνοντα φτώχεια από τα άλλα και εξαγοντά την, διότι μιλάμε για πολιτική συνοχή. Ε, αυτό δεν μπορεί να τα ε, κουμπίσει κανείς ή τα κονδύλια των μεταφορών έχουν στοχευτεί για τις μεταφορές και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές. Αυτά. Είχατε κάποια μικροσχόλια, αλλά σας έχω γράψει ένα mail. Τι εννοείται διεθνείς οργανισμοί. Χρειάζονται την έγκριση των κρατών μελών. Από πού και ως πού. Δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου, κύριε Τελίτσκα, για δύο λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα έχουμε ήδη συζητήσει, γι' αυτό θα είμαι σύντομο. Και ε, επιπλέον τον όσον είπε ο κύριος Μαρινέσκου. Σημειώνουμε αυτό που μας λέτε, ότι είναι μια πολύ ξεκάθαρη πρόταση για να λειτουργήσει και να... Και αυτό είναι κάτι που το εκτιμούμε, αλλά δεν είναι σίγουρα τέλεια. Ε, επιδιώκαμε την απλούστευση, να ενθαρρύνουμε τα πράγματα που πηγαίνουν καλά, να δούμε πού δεν πάνε καλά και που υπάρχουν δυσκολίες και κενά για την ε, ψηφιοποίηση το θέμα της κινητικότητας, ε, της ιδιωτικής κινητικότητας ήδη το έθιξε ο κ. Μανέσκου. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και ότι δεν ξέρουμε. Ε, για 6,5 δις μου φαίνεται λίγο ε, άσκοπο σχόλιο. Πρέπει να ξέρουμε και να το αξιοποιήσουμε και νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε. Θα πρέπει να τα πλουστεύσουμε εδώ λίγο τα πράγματα ε, και να είναι σαφές εδώ, αλλά θα πρέπει η αισθητική συνιστόσα να βασιστεί στα υπάρχοντα δίκτυα TNT και στις υπάρχουσες μελέτες σκοπιμότητας, τα έργα και την υλοποίηση. Ο κύριος Μαρινέσκου τόνισε το θέμα και το 30-50 για τη συνοχή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιζητήσουμε κάποια εξισορρόπηση μεταξύ της διάστασης ανταγωνισμού και μετά Ε, και όπως είπε και ο κ. Μαρινέσκου, γιατί κάποια κράτη-μέλη δυσκολεύονται να συγχρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα, ας πούμε οι χώρες των Βαλκανίων. Από την άλλη υπάρχουν άλλες χώρες συνοχής που θα χρηματοδοτούν κάτι άλλο και θα αποκαλέσει κάποιο το ένα θέμα του ανταγωνισμού κτλ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά μιλήσατε για την ε, αναλογία 60-40. Δεν μου φαίνεται και πολύ καλή ιδέα. Είναι ένα παράδειγμα του που μπορούμε να επιδιώξουμε απλούστευση, για το blending, για, την, ε, για το συνδυασμό και την ανάμειξη. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι εδώ. Αλλά πρέπει να μας απασχολήσει ότι είναι και εφικτό. Έχω και άλλες παρατηρήσεις, αλλά καμία δεν είναι τελείως άγνωστη. Νομίζω ότι και με τον κύριο Μαρινέσκου και με την κυρία Βιρκούνεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά σε μια ομάδα. Είναι πολλά αυτά θα πρέπει να χτενίσουμε αλλά η πρώτη μετάφραση νομίζω θα είναι ήδη έτοιμη στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Πρόεδρο. Και τώρα οι βουλευτέ μας. Για ένα λεπτό, κυρία Ντεμόντε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα νέα στοιχεία για το τούνελ του Μπρένερο και για τη συνεργειακή σύνδεση της ταιριέ της με την μπάτσα και για την στρατηγική κινητικότητα. Τι στρατηγικές έχετε σκεφτεί πού θα παρέμβουμε σε κάποιο είδους ε, γέφυρες για δυσυνοριακές διασυνδέσεις. Ευχαριστούμε κύριο Ζήλε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κατά πρώτον. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που θα παρεμβουμε σε καποιο ειδους γεφυρες για συνοριακές διασυνδεσεις ευχαριστουμε κυριο ζηλε για ευχαριστω κατα πρωτον ειμαι πολυ ικανοποιημενο με αυτα που προτεινει η Κομισιόν. Ίσως για το Ταμείο συνοχή έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά ο ανταγωνισμός για το κομμάτι αυτό το προβλησμό είναι πολύ σημαντικός. Θα ήθελα να βλέπαμε ότι, όμως ότι υπάρχουν κάποιες αδικίες γιατί υπάρχουν ε, χώρες, ε, περιοχές ψηλής και χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού. Οπότε τα κόστη για τις χώρες που έχουν χαμηλή ε, πυκνότητα ε, είναι υψηλότερα. Πρέπει όμως να ολοκληρωθούν τα project που έχουν ήδη ξεκινήσει γιατί αλλιώς πώς θα εξηγήσουμε πώς ξοδέψαμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και τελικά δεν ε, ολοκληρώσαμε τέτοιου είδου μεγάλα δίκτυα τα επόμενα 6-7 χρόνια. Αυτά που ξεκίνησαν θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν. Κύριε Κράμερ, θέλετε το λόγο. Σας ευχαριστώ ε, για αυτή την παρουσίαση και χαίρομαι για το ότι έχετε δώσει ε, έμφαση στο cross-border, στο διασυνοριακό, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε για να μην πούμε ότι και οι νέες και οι παλιές προτεραιότητες είναι ειδήσεις γιατί βέβαια αν το πούμε αυτό, το ουσιαστικά θα πάνε όλα τα κονδύλια στις παλιές και τίποτα στις καινούριες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό έχετε δίκιο αλλά σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση και το κενό που υπάρχει εκεί. Ε, δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, είχαμε την σύνδεση Μπερλίν-Στετίν, 30 χιλιόμετρων, έγιναν συζητήσει ξανά και ξανά, αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν δείχνει ενδιαφέρον. Ή δεν την ενδιαφέρει καθόλου, για παράδειγμα, η επανασύνδεση με την Πολωνία. Άρα, σε αυτέ τι περιπτώσει, τι είδου δυνατότητε έχει η Επιτροπή προκειμένου να επιβάλλει, αν θέλετε, το εισαγωγικό κάποιε συνδέσει ακόμα και αν τα κράτη-μέλη δεν τις υποστηρίζουν. Δηλαδή μπορούν, για παράδειγμα, ε, να υποστηρίξετε κάτι τέτοιο. Υπήρξε, για παράδειγμα, μία σύνδεση και μετά από το σύγχρονο παραπέτασμα, αλλά μεταξύ Γερμανία και Πολωνία, αλλά μετά από πέντε, ή μάλλον εδώ και πέντε χρόνια Πολωνία δεν ε, θέλει πλέον συνεχίσετε αυτή η σύνδεση. Οπότε θα πρέπει, ε, ενώ έχει επανασταθεί αυτή η σύνδεση, η Πολωνία δεν θέλει να το κάνει γιατί να συνεχίσει τη σύνδεση γιατί είναι τεχνικά δύσκολη. Οπότε δεν πρέπει να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Αμάτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ναι, κάποιε παρατηρήσει κυρίω για τον προγραμματισμό 2014-2020. Έχουμε απορίε σε σχέση με τα κονδύλια του προπολογισμού. Κυρίω για τα ποσά για τι μεταφορέ. Προτείνονται 30 δι επιπλέον, 30,5 δι, και 6,5 για τη στρατηγική κινητικότητα. Θα συμφωνήσω με τι απορίε των συναδέλφων, διότι δεν γνωρίζουμε, δεν είναι σαφεί οι προποθέσει και οι προτεραιότητε. Έχουμε λοιπόν σοβαρέ αμφιβολίε για την ανάγκη να δαπανηθούν αυτά τα δι για την θεατρική κινητικότητα. 11,3 για τι υποδομέ των υποπροσχώρηση χωρών και συνοχή και 18 για το ΣΕΦ συνολικά ουσιαστικά ε, τόσο για την άμυνα, τόσο για τη συνοχή. Μένουν 12,8 για την Ευρώπη των 27 ε, ε, κρατών, το 42%. Εντάξει, θέλουμε τα κονδύλια της συνοχής. Εγώ είμαι πλήρες μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς Θεού. Αλλά όλα αυτά, όχι για να ευβληθούν... Να ωφεληθούν μάλλον και οι εξόχους από και τις περιοχές της συνοχής, όπως ο νότος της Ιταλίας. Και η Ιταλία δεν έχει μπορέσει να αξιοποιήσει τα κονδύλια για τη διασύνδεση, τη διασυνοριακή, μέσα στην Ιταλία και στα σύνορα προ το βορρά. Ευχαριστούμε κυρία Μάτο, Νταμάτο. Θα σας αφήσω να απαντήσετε αγγλικά κύριε Ρόιτερς. Ευχαριστούμε τους Γερμενείς. Ε, ναι, είδαμε ότι μας κάνατε νόημα και θα συνεχίσουμε για λίγα λεπτά στα αγγλικά. Ε, όπως σας είχαμε πει, εμείς δεν μπορούμε να σας παραχωρήσουμε υπέρβαση του ωραρίου σήμερα στη σημερινή συνεδρία. Ευχαριστούμε. Well. Uh, ladies and gentlemen, thank you for, for the uh, questions that were raised. I think I will uh, take a few uh, themes uh, briefly